Ich bitte Platz zu nehmen. Καλό καθίστε κυρίες και κύριοι. Θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Αντίθετα όμως με μένα που δεν ήμουν το πρωί, οι άλλοι ήσασταν το πρωί. Σας ευχαριστώ λοιπόν που με εκλέξατε παρόλα αυτά, Πρόεδρο. Σας υπόσχομαι πως ε, θα προσπαθήσω να συνεργαστώ στενά με την Επιτροπή και πρέπει να σκεφτούμε γρήγορα ποιες ε, πολιτικές προτεραιότητες θα θέσουμε ε, έτσι ώστε προς λύπη της Κομισιόν και της Υπηρεσίας Εξωτερικών Υποθέσεων να χαράξουμε σκληρές στρατηγικές. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Θα πρέπει να εργαστούμε σκληρά τις επόμενες εβδομάδες. Εγώ λοιπόν τη χαρά τώρα να καλωσορίζω τον Επίτροπο ε, Διεύρυνσης και Πολιτικής Γειτονίας, τον κύριο Φίλε, ο οποίος ε, θα μας κάνει μια παρουσίαση, αλλά πριν από αυτό νομίζω θα λάβει τον λόγο ο συντονιστής της συζήτησης, ο Νάτσο. Ευχαριστώ Ελμάρ και εγώ θα ήθελα να υποδεχθώ τον ε, Επίτροπο Φούλε ε, αλλά και τον Γενικό Γραμματέα της ΕΑΣ ε, Πιέρ Δημό Σήμερα το πρωί ο πρέσβης Τέιλορ ε, έλεγε ότι εμείς από ευρωπαϊκή πλευράς ε, κάναμε κάποια σφάλματα και δημιουργήσαμε μια έλλειψη αξιοπιστίας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να κάνουμε όμως μια σαφή μια, προσπάθεια προκειμένου να καταδείξουμε ότι δεν, ε, τα σφάλματά μας δεν ήταν ηθελημένα. Τώρα γίνανε κάποιες εκλογές όπως ξέρετε σε πολλές ε, χώρες. Ε, μεταξύ επίκυνται νέε εκλογές στην Αλγερία. Νομίζω πως δόθηκε απάντηση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της κοινή ανακοίνωσης της υπηρεσίας κοινή δράσης που οποία ε, ζητούσε να υποστηρίξουμε αυτές τις διαδικασίες τις μεταβατικές αλλά και τις προσπάθειες οικονομικής ανάπτυξης αλλά παράλληλα και την περιφερειακή ανάπτυξη και συνεργασία ε, με τους απαραίτητους μηχανισμούς προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αυτή η κατάσταση. Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να ζω τον κύριο Φίλε, σήμερα το πρωί ήδη συζητήθηκε το θέμα, να το ζητήσω κάτι σχετικά με τις προϋποθέσεις, με τους όρους, ε, με την αιρεσιμότητα. Να καθορίσουμε λοιπόν κάποια κριτήρια ε, αναφορικά με το τι, πώς διευθετήθηκε αυτή η απάντηση και πώς θα διαμορφωθεί σε σχέση με το μέλλον και τις εξελίξεις. Ε, μια που έχουμε ανάμεσα με τον Δημού, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το νέο πολιτικό σκηνικό το οποίο προέκυψε από τις εκλογές, από τις κάλπες και να δούμε τι η μέτρο Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ε, προωθήσει τις σχέσεις μας ε, με τις κυβερνήσεις ε, οι οποίες προκύπτουν μετά από τις εξελίξεις στις χώρες αυτές. Ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών των ο κ. Μπέκερ έλεγε πως η διπλωματία είναι μια δραστηριότητα την οποία θα πρέπει να καλλιεργούμε σε κάποιο εντύνη μέτρο όπως και η Κυπουρική. Θα πρέπει λοιπόν να τη φροντίζουμε, να την ποτίζουμε, να την κλαδεύουμε κλπ. πράγματα όμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα, δεν είναι όπως ήταν στο παρελθόν ότι σηκώναμε το τηλέφωνο και ε, ζητούσαμε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο με το οποίο θα ερχόμαστε σε επαφή. Τα πράγματα τώρα αλλάζουν ε, και γι' αυτό θα χρειαστεί ο πλευράς μας ε, να καταβληθεί σημαντική προσπάθεια. Θα πρέπει λοιπόν ε, οι υπεύθυνοι να αναλάβουν την κατάλληλη δράση και θα θέλω να ζητήσω από τον Επίτροπο κύριο Φίλε να μας κάνει μια παρουσίαση το χρόνο που του έχει δοθεί και να ακούσουμε μετά τις ε, θέσεις και τα σχόλια των μιλών του Ευρωκοινοβουλίου αλλά και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ευχαριστώ. Thank you, uh, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και συγχαρητήρια. Κυρίε και κύριοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων, σας ευχαριστώ που με καλέσατε σήμερα εδώ ε, και για το ότι επίσης προσκαλέσατε τόσους πολλούς ε, εθνικούς βουλευτές. Ήδη έχει περάσει πάνω από ένα έτος από τις πρώτες διαμαρτυρίες ε, της Αραβικής ε, Άνοιξης που ξεκίνησαν μια σειρά γεγονότων η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Είδαμε τους λαούς της περιοχής που εξέφρασαν την επιθυμία τους για ένα καλύτερο μέλλον, για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και για μια τη ζωή με αξιοπρέπεια και τους αυτούς τους και τις μελλοντικέ γενναίες. Σε λίγες χώρες είχαμε πραγματικά γνήσια και εντυπωσιακή πρόοδο. Ιδιαίτερα αναφέρομαι στην Τινησία αλλά και το Μαρόκο. Σε άλλες ξεκίνησαν μεταρρυθμίσεις αλλά ακόμα πρέπει να γίνουν πολλά για να εκπληρωθούν οι φιλοδοξίες του λαού. Κυρίως εννοώ την Αλγερία όπου έχουν γίνει πολλές μεταρρυθμίσεις και καλείται η Ευρωπαϊκή Ένωση να τις υποστηρίξει στο πλαίσιο ενός νέου σχεδίου δράσης και να στείλει ένα σαφές μήνυμα στήριξης και ενδιαφέροντος για την πολιτική γειτονία που υπάρχει και από πλευράς Αλγερίας. Σε άλλες χώρες όμως η κατεύθυνση δεν έχει πάει στην σωστή κατεύθυνση. Συνολικά είναι σαφές πως η κατεύθυνση του δημοκρατισμού θα είναι η διαδικασία αυτή μακρά. Θα υπάρξουν βήματα προς τα πίσω και απογοητεύσεις, αλλά είμαι σίγουρος πως έχουν πλέον απελευθερωθεί ισχυρέ δημοκρατικές δυνάμεις και έχουν αποκτήσει εξουσία πολίτε πολίτες. Πριν από λίγους μήνες ήρθα εδώ πέρα και σας παρουσίασα την αξιολόγησή μου για τα γεγονότα που εκτελήσονταν. Τότε αναγνώρισα πως η πολιτική μας στην περιοχή δεν ήταν πάντα η σωστή. 11 μήνες αργότερα πρέπει να παραδεχτώ πως εξακολουθώ να ε, θεωρώ πως μπορούμε όλοι να αποφεληθούμε από μια συνεχή επαφή με την πραγματικότητα και έλεγχο του εάν η πολιτική μας είναι στο ύψος των ιστορικών προκλήσεων. Γνωρίζω πως συνεχώς αγωνιζόμαστε από κοινού, κύριε Πρόεδρε, για να διατηρήσουμε τις αξίες και τα συμφέροντά μας όσο το δυνατόν πιο κοντά. Στη σχέση μας με τους νότιους γειτονές μας είναι φανερό πως δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στις παλαιές ημέρες όπου αντιμετωπίζαμε ήπια τα καθεστώτα τα αυταρχικά. Τώρα πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να δρανεί ενώ η ιστορία προχωράει μπροστά. Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να υπενθυμίσω τους γενικούς μας στόχους πριν σας ενημερώσω για την εφαρμογή, την εφαρμογή τους και τις προκλήσεις ε, του μέλλοντος. Ε, πρώτος μας στόχος είναι να υποστηρίξουμε τους εταίρους μας οι οποίοι κάνουν μεταρρυθμίσει στην κατεύθυνση της βαθιάς δημοκρατίας του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για να υπάρχει διαρκής και γνήσια ευμερία και σταθερότητα, όχι σταθερότητα που προστατεύει ε, αυταρχικά καθεστώτα, αλλά σταθερότητα η οποία διασφαλίζει πως υπάρχει αρμονική και αξιοπρεπής ανάπτυξη των εταίρων μας και των λαών τους. Δεύτερο στόχος μας είναι να υπάρξει μια συνεργασία με τις κοινωνίες παράλληλα με τη συνεργασία των κυβερνήσεων. Η προσέγγιση μας βασίζεται σε δύο βασικές αρχές για περισσότερη και αμοιβαία λογοδοσία. Όσον αφορά το πρώτο θα σας πω σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια πώς σκοπεύουμε να ε, το εφαρμόσουμε ε, αυτό. Είναι σαφές πώς εξακολουθούμε να έχουμε μια προσέγγιση η οποία βασίζεται σε μια αιρεσιμότητα θετική και μια ευελιξία η οποία θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προσαρμόσει τα κίνητρά της στις προκλήσεις και ευκαιρίες οι οποίες αλλάζουν. Και βεβαίως, αναμένω τη συζήτηση αυτή μαζί σας και με άλλους ενδιαφερομένους σε ευθετότερο χρόνο κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα τώρα να τονίσω κάποια επιτεύγματα των τριών στόχων μας, ε, των τριών πτυχών αυτών, ε, που είναι τα λεγόμενα χρήματα, κινητικότητα και αγορές. Όσον αφορά τα χρήματα, πρώτα απ' όλα διαθέσαμε ένα δισεκατομμύριο παραπάνω το 2011, το οποίο προστίθεται στα 7,5 δισεκατομμύρια που υπήρχαν ήδη. Επίσης υπάρχει ένα νέο πρόγραμμα ονόματι Spring, ε, που είναι ένα αρκτικό λεξο βεβαίως, το οποίο καταλήγει στο ε, ακρονίμιο Spring, δηλαδή Άνοιξη. Πρόκειται για επιπλέον 350 εκατομμύρια για το 2011 και 2012 που στηρίζει τις χώρες αυτές οι οποίες εδρεώνουν τις μεταρρυθμίσεις. Πέρα από αυτά τα κονδύλια, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα διαθέσει κονδύλια και μάλιστα αυτά αυξήθηκαν κατά ένα δισεκατομμύριο. Η εντολή δανεισμού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης επίσης επεκτάθηκε και άρα θα υπάρχουν ακόμα 2,5 δισεκατομμύρια διαθέσιμα το έτος. Σημαντικό σημείο επίσης προσοχής ήταν η ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών. Ξεκίνησε λοιπόν το μέσο κοινωνίας των πολιτών να λειτουργεί τον περασμένο Σεπτέμβριο και συνεχίζεται με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία. Η Κομισιόν επίσης ανανέωσε και αύξησε την χρηματοδότησή της στο Ίδρυμα Αναλίντ. Και τέλος, ενισχύσαμε τη συνεργασία μας με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Την προηγούμενη εβδομάδα μόλις ε, συμφωνήσαμε σε ένα νέο πρόγραμμα 4,8 εκατομμυρίων ευρώ για να ενισχύσουμε την πολιτική και οικονομική μεταρρύθμιση στην περιοχή της νότιας γειτονίας μας, ξεκινώντας από την Τινησία και το Μαρόκο. Χρησιμοποιώντας λοιπόν όλη την προσθέμενη αξία και την πείρα του Συμβουλίου της Ευρώπης όσον αφορά την πολιτική γειτονία και την ε, εταιρική σχέση για τις μεταρρυθμίσεις και την δημοκρατία που έχουν ήδη με την Τινησία και το Μαρόκο και θα προσπαθήσουμε να το επεκτείνουμε και με άλλους ε, εταίρους στο Νότο. Θα χρειαστούμε όμως και άλλα. Πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών με τις ε, χώρες αυτές ε, στο πλαίσιο των προγραμμάτων μας. Επίσης πρέπει να υπάρξει ένας πιο τακτικός και δομημένος διάλογος με την κοινωνία των πολιτών επί τόπου για να επωφεληθούμε σε χρόνο άμεσο από την εμπειρία τους και βεβαίως να ενημερώσουμε καλύτερα για τις δραστηριότητες μας. Η αύξηση της κινητικότητας και των επαφών μεταξύ των λαών βεβαίως είναι κρίσιμη σημασία σε αν αυτό το οποίο λέει η Ευρώπη πως θέλει μια πραγματική εταιρική σχέση με τους γειτονές μας στη Μεσόγειο είναι κάτι το οποίο παίρνουμε σοβαρά χαίρομαι για το ότι οι εταιρικέ σχέσεις κινητικότητας έχουν ξεκινήσει με την την Ισία και το Μαρόκο τον Οκτώβριο του 2011 και ελπίζω πως θα υπογραφούν υπό την Προεδρία της Δανίας. Οι συνεργασίες αυτές θα βοηθήσουν να αναπτύξουμε συνολική και ισορροπημένη συνεργασία στην ε, διαχείριση της ε, νόμιμης ε, και παράνομης μετανάστευσης, της επανεισδοχής, των θεωρήσεων, της διεθνούς προστασίας, και ζημάτων ασφάλειας και συνόρων. Επίσης, 740 επιπλέον υποτροφίες Εράσμους Μούντους για ανταλλαγέ μεταξύ πανεπιστημίων με την ε, νότια όχθη της Μεσογείου χρηματοδοτήθηκαν για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Άλλα 80 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στις χώρες ε, της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας το 2012 και 2013 για τον ίδιο σκοπό. Τα μέτρα αυτά θα προωθήσουν την αμοιβαία κατανόηση. Επίσης θα βοηθήσουν τους γείτονές μας στο να αναπτύξουν τις δεξιότητες και την εμπειρία που χρειάζονται για να είναι επιτυχής η μετάβασή τους. Τέλος, οι αγορές. Οι εντολές για την ανάπτυξη συνολικών συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου με την Αίγυπτο, την Ισία, Μαρόκο και η Ορδανία εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 14 Δεκεμβρίου. Αυτές θα διευκολύνουν σταδιακή και βαθύτερη οικονομική ενσωμάτωση με την εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά οι συμφωνίες αυτές βεβαίως θα τεθούν σε ισχύ σε κάποιο βάθος χρόνου. Ταυτόχρονα εξετάζουμε εμπορικά μέτρα τα οποία μπορούν να εισαχθούν γρήγορα και τα οποία θα είναι αμοιβαίως εποφελή. Η, η Συμφωνία Απελευθέρωσης Αγροτικών Προϊόντων με το Μαρόκο είναι ένα τέτοιο μέτρο και ελπίζω θέλω να το τονίσω αυτό, πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δώσει τη σύμφωνη γνώμη του στην Ολομέλεια του Φεβρουαρίου. Ελπίζουμε επίσης να συναυθεί ανάλογη συμφωνία με την Τινησία. Τέλος, πέρα από αυτά τα τρία σημεία που ανέφερα, δραστηριοποιούμαστε σε κάποια άλλα τομεακά ζητήματα, μεταφορές, ενέργεια και τεχνολογία της ε, πληροφορίας. Σε όλα αυτά εντείνουμε τη συνεργασία μας με τους γείτονές μας προς Νότον. Θα ήθελα να τονίσω, κύριε Πρόεδρε, πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωριστεί ως βασικός εταίρος για την οργάνωση και την παρακολούθηση των δημοκρατικών εκλογών στην περιοχή. Η βοήθειά μας και η αποστολή μας στην ε, Ισία... Ε, ήταν κάτι το οποίο εκτιμήθηκε δεόντως και είμαι υπερήφανος για το ότι οι αρχές της Αλγερίας μας προσκάλεσαν μεταξύ άλλων διεθνών οργανισμών να παρατηρήσουμε τις εκλογές οι οποίες θα διεξαχθούν. Επίσης μας ζητήθηκε να υποστηρίξουμε με την εμπειρογνωμοσύνη μας το Μαρόκο και τους εθνικούς παρατηρητές των εκλογών στην Αίγυπτο. Καθώς λοιπόν κοιτάμε το μέλλον βλέπουμε πως για κάθε χώρα η μετάβαση είναι διαφορετική. Άρα πρέπει να υπάρξει ένας μοναδικός διάλογος για να υπάρχει μια συνολική και πλήρη στήριξη αυτής της διαδικασίας. Αυτός ο διάλογος πρέπει να συμπεριλάβει όλους τους εταίρους. Κυβέρνηση, επιχειρήσεις, ε, κοινωνία των πολιτών κτλ. Μόνο τότε θα έχουμε την απαραίτητη αυτή ε, αντίδραση των συμμελιτών μας για να μπορούμε να προσαρμόσουμε ανάλογα την πολιτική μας η πολιτική στήριξη των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στη νότια γειτονιά μας είναι κάτι το δεδομένο. Πρέπει λοιπόν τώρα να φροντίσουμε πως όλα αυτά θα γίνουν με τρόπο έγκαιρο και στοχευμένο επιτόπου. Και άρα ε, στο πλαίσιο αυτό η ομάδα εργασίας που συνέστησε η κάθε άστον ή του εκπρόσωπο και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει να παίξει ένα ρόλο κλειδί ειδικά όσον αφορά το συντονισμό της αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των κρατών μελών της και των Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών ε, Οργάνων. Πρόκειται λοιπόν για μια διαδικασία μακροπρόθεσμη. Την τελευταία φορά που επισκέφθηκα την περιοχή μου είπαν πως η επιτυχημένη μετάβαση δεν είναι κάτι το οποίο θα μετρήσουμε στον πρώτο γύρο των δημοκρατικών εκλογών, αλλά στον δεύτερο, τρίτο και τέταρτο. Πρέπει λοιπόν να αναπτύξουμε σχέσεις με την νέα ηγεσία και να συνεργαστούμε για να έχει βαρά θεμέλια η δημοκρατία και η ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την εμπειρία 100 μελών που πέρασαν μια παρόμοια διαδικασία και μπορεί επίσης να προσφέρει την εμπειρία της περιφερειακής ολοκλήρωσης. Γνωρίζουμε πως η μεγαλύτερη οικονομική ολοκλήρωση και συνεργασία μεταξύ των χωρών του Μαγκρέβ δεν θα αυξήσει μόνο το ΑΕΠ τους κατά 2% αλλά θα αποτελέσει καταλήτη για την εδραίωση της διαδικασίας αυτής δημοκρατικού μετασχηματισμού. Στο πλαίσιο αυτό με ενθαρρύνουν οι επαφές μεταξύ Μαρόκου και Αλγερίας και ελπίζω η Ένωση για τη Μεσόγειο να μπορέσει να λειτουργεί, να αρχίσει να λειτουργεί και να προσθέσει περαιτέρω αξία με το να βρίσκει ποια είναι τα κατάλληλα εκείνα έργα που πρέπει να ενισχυθούν, που θα αυξήσουν την αλληλεγγύη στη Μεσόγειο. Και δεν θα πρέπει να φοβόμαστε το αποτέλεσμα δημοκρατικών εκλογών. Πρέπει να είμαστε σε επαφή με τους εταίρους μας και να τους κρίνουμε με βάση τα γεγονότα και το πώς σέβονται τις διεθνείς τους δεσμεύσεις. Την προηγούμενη εβδομάδα ημουν στο Μαρόκο οπου συνάντησα τον νέο Πρωθυπουργό, ο οποίος επιβεβαίωσε πως είναι πρόθεση της κυβέρνησής του να βελτιώσει τις εμελιώδεις ελευθερίες και την διοίκηση και επίσης την εταιρική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και χαίρομαι για το ότι ο Πρωθυπουργό τη Τινησία την ερχόμενη εβδομάδα σκοπεύει να μα επισκεφθεί για να δείξει το πόσο θέλει η κυβέρνησή του να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνοντα, θα ήθελα να πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μεγάλη ευθύνη να παρακολουθήσει αυτή τη διαδικασία μετασχηματισμού, όχι μόνο συνεργαζόμενο χέρι με χέρι με τα άλλα θεσμικά όργανα τη Ένωση και να υποστηρίξει τις προτάσεις Κομισιόν για να δώσουμε μεγαλύτερο βάρος και οικονομικούς πόρους στη γειτονιά μας, αλλά συνεργαζόμενο και με τα κοινοβούλια των εταίρων μας με το να ταξιδεύει στην περιοχή αυτή και να αναγνωρίσει τον ρόλο αυτών οι οποίοι φέρνουν την αλλαγή. Και είμαι σίγουρος πως συνεργαζόμενοι μαζί σας μπορούμε να υποστηρίξουμε μία μόνιμη μετάβαση και τον εκδημοκρατισμό. Να με λοιπόν τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Thank you, Commissioner. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Πριν δώσω το λόγο στον επόμενο μιλητή θέλω να τονίσω ότι το πρωί ο ε, πρέσβης Τέιλορ είπε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες ανεγνώρισαν λάθη αλλά και εμείς στην Ένωση πράξαμε λάθη. Ο κύριος Ρομπιμόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα μακρηγορήσω. Θα σας κάνω μερικές παρατηρήσεις ως προς το τι συμβαίνει πολιτικά αυτή τη στιγμή στις διάφορες χώρες που, όπου σημειώνονται τα γεγονότα αυτά που ονομάζουμε Αραβική Άνοιξη. Και αυτό διότι νομίζω ότι ο Επίτροπος Φιούλε τα είπε όλα και μου έμειναν λίγα να προσθέσω. Καλύτερα λοιπόν να σας κάνω μερικά σχόλια για να δούμε τι συμβαίνει στις χώρες αυτές και να καταλήξουμε σε μερικές κατευθυντήριες γραμμές που να εφαρμόσουμε στην ανταπόκριση που θέλουμε να δώσουμε στα γεγονότα αυτά. Πρώτον, αν θέλουμε να καταλάβουμε τι πράγματι συμβαίνει, πρέπει να είμαστε ακριβείς και να καταλάβουμε ότι η κατάσταση σε κάθε μια από αυτές τις χώρες είναι διαφορετική από τον άλλον και ότι επομένως αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε διότι πολλές από... οι χώρες αυτές δεν έχουν όλες την ίδια πολιτική ιστορία και παράδοση ακόμη και αν μιλάμε για μουσουλμανικά κόμματα Ισλαμικά κόμματα δεν πρέπει να συγχαίουμε το Εναχντά στην Τινησία με την ε, μουσουλμανική αδελφότητα στην Αίγυπτο. Άλλες παραδόσεις έχουν. Κάποτε οι ηγέτες της Εναχντά είχαν εισέλθει σε μια πολύ μεγάλη και μακροχρόνια διαμάχη με τη μουσουλμανική αδελφότητα στο Σουδάν. Η διαμάχη αυτή και η συζήτηση αφορούσε ακριβώς το τι είναι ακριβώ το πολιτικό Ισλάμ και ποια σχέση έχει με τη δημοκρατία, το ρόλο που μπορεί και πρέπει να παίζει το Κοράνι στην πολιτική ζωή. Δεν αρχίζουμε λοιπόν από το μηδέν. Ήδη έχουν συζητηθεί αυτά τα πράγματα πολλές φορές για πολύ καιρό. Αν θέλουμε να συνοψίσουμε την κατάσταση θα λέγαμε ότι πρώτον βλέπουμε ότι υπάρχουν χώρες όπου η εκλογική διαδικασία έγινε, πραγματοποιήθηκε και ήδη συστήθηκαν καινούργιες κυβερνήσεις, η Τινησία και το Μαρόκο. Έπειτα υπάρχουν χώρες όπου είχαν γίνει εκλογές, όπως στην Αίγυπτο, αλλά δεν έχει ακόμα συσταθεί νέα κυβέρνηση. είναι η μετάβαση δεν είναι πολύ ομαλή. Η σχέση στρατού και κοινωνίας πρέπει να διευθετηθούν για να μπορέσει πλήρως ο στρατός να αποσυρθεί από την πολιτική ζωή και να δώσει την εξουσία στην πολιτική κυβέρνηση. Συνεχίζονται οι συνεννοήσεις και μπορεί να χρειαστεί κάποιος χρόνος. Και επίσης υπάρχει μια συνταγματική διαδικασία. Τρίτον, υπάρχουν χώρες όπου η αλλαγή του καθεστώτος υπήρξε, αλλά δεν έχουν ακόμη τουλάχιστον διοργανωθεί εκλογές η Εμένοι, η Λιβύη και κάθε μέρα βλέπουμε ότι η κατάσταση εκεί παραμένει ασταθής, αν και δεν υπάρχουν τα ίδια γεγονότα και η ίδια αστάθεια που παρατηρείται στη Συρία ή και στο Μπαχρέιν που είναι ίσως η επόμενη κατηγορία χωρών που ζουν ακόμη μεγάλη αστάθεια. Τέλος υπάρχει και μια κατηγορία όπου αναμένονται αλλαγές, έχουν ανακοινωθεί, αλλά πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Η Ορδανία, Αλγερία, όπου προβλέπονται εκλογές και μα θύμισε ο Στέφεν ότι θα υπάρξει και εποπτεία εκεί αλλά και εκεί πρέπει μάλλον να πούμε ότι θα γίνει μια σημαντική αλλαγή. Αυτή είναι η πραγματικότητα που παρατηρούμε και επομένως επαναλαμβάνω ότι όταν μιλάμε για την Αίγυπτο ή την Τινησία πρέπει να γνωρίζουμε τις διαφορές αυτές. Μια τελευταία παρατήρηση. Όλοι εκπλήσονται από το ρόλο που παίζει η Τινησία, από τον τρόπο με τον οποίο γίνανε τα πράγματα μέχρι τώρα. Αλλά μην ξεχνάτε ότι υπάρχει μεγάλη ιστορία στην Τινησία που μπορεί να την έχουν μερικοί ξεχάσει. Πριν από τον Μπεναλή υπήρχε ο Μπουργκίμπα. Και όταν έγινε ανεξάρτητη η Τινησία, ο Μπουργκίμπα θεωρούνταν από πολλούς πολιτικούς παρατηρητές ως ηγέτης πολύ παρόμοιος με τις ιδέες του Ατατούρκ. Και ένας από τους λόγους για τους οποίους βλέπουμε τι γίνεται στην Τινησία, γίνονται αυτά που γίνονται στην Τινησία, είναι ότι οργανώνονται δημόσιες συζητήσεις και αυτό οφείλεται εν πολλής στο ότι υπήρξε αυτή η προϊστορία η ελευθερία των γυναικών, η πολιτική συζήτηση, η κοσμική κοινωνία για αρκετό καιρό. Βέβαια έχουμε παρατηρήσει και πολλές ελλείψεις στην Τινησία από την ανεξαρτησία και μετά, αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχει αυτή η προϊστορία και αυτή η μνήμη σε ό,τι συζητιέται αυτή τη στιγμή στην Τινησία. Αυτή ήταν η πρώτη μου παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση, η δική μας παρέμβαση στη χώρα αυτή πρέπει να είναι ακριβώς προσαρμοσμένη στις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή εκείνη. Όπως και σε κάθε χώρα βέβαια. Και νομίζω ότι φάση με τη φάση πρέπει να προσαρμοζόμαστε στα γεγονότα που ε- όπως εξελίσσονται. Καταρχάς προσφέραμε στήριξη στην εκλογική διαδικασία και στη συνταγματική διαδικασία στην Τινησία Προτείναμε επίσης και στην Αίγυπτο ανάλογη βοήθεια και συνεργαστήκαμε στενά και με την κοινωνία των πολιτών στη Λιβύη, τουλάχιστον στη Βενγκάζη. Δεύτερη φάση. Προσφέραμε βοήθεια στις δυνατότητες οικοδόμησης της κοινωνίας των πολιτών και εδώ χρησιμοποιούμε ό,τι εργαλεία διαθέτουμε, ιδιαίτερα το εργαλείο σταθερότητας, αλλά καθώς ελπίζουμε να ιδρύσουμε το European Endowment for Democracy, Ελπίζουμε ότι και αυτό θα βοηθήσει στην εξέλιξη των πραγμάτων. Τρίτη φάση, όταν μας το ζήτησαν, θελήσαμε να αντιμετωπίσουμε τα πιο επίγοντα προβλήματα. Οι μεταβατικές αρχές δηλαδή μας ζήτησαν, η, Λιβύη η Λιβύη ζήτησε πολύ απλά να τους βοηθήσουμε για τρία θέματα. Τους συνοριακούς ελέγχους, την ασφάλεια και ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση των επικοινωνιών και των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τις αρχές εκεί, διότι ένα χαρακτηριστικό που είναι κοινό είναι ότι πάντοτε μας θυμίζουν την ανεξαρτησία και κυριαρχία τους. Εμείς δεν μπορούμε ούτε για ένα λεπτό να σκεφτούμε ότι θα πάμε να επιβάλλουμε αυτό που θεωρούμε σωστό. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα της κατάστασης που αντιμετωπίζουμε. Η τωρινή κυβέρνηση στη Λιβύη θεωρεί τον εαυτό της ως προσωρινή κυβέρνηση. Θα οργανωθούν εκλογές πριν λέει το καλοκαίρι. Και θέλουμε να αναγνωρίσουμε το βαθμό στον οποίο ζήτησαν βοήθεια. Δεν θέλουν με κανένα τρόπο να επιβληθεί στους ε, επόμενους, στην επόμενη κυβέρνηση η δική μας λύση. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε με πολύ προσοχή μαζί τους και να δούμε μέχρι ποιο σημείο μπορούμε να πάμε χωρίς να θεωρήσουν οι αρχές αυτές ότι επιβάλλεται μια λύση για τους διαδόχους τους. Τέταρτη φάση που αφορά όλες τις ιδέες και προτάσεις που σας ανέφερε και ο Επίτροπος Σούλε προηγουμένως είναι η πιο μακροπρόθεσμη δράση που μπορούμε να αναλάβουμε εμπορική, εκπαιδευτική, επενδυτική, μεταναστευτική. Μας είπε ο Επίτροπος Φίλε προηγουμένως ότι όπως σας είπε και ο Μπερναρδίνο Λεόν το πρωί ότι έχουμε μια ειδική ομάδα επιτροπή για την Τινησία και το ίδιο θα κάνουμε για την Ιορδανία. Η ΔΕ Λέδη Άστον θα συμμετάσχει και θα πάει στην Ιορδανία και θα ζητήσει από μερικούς από εσά να συμμετάσχετε και εσείς σε επίσκεψη τουλάχιστον στην Ειδική Επιτροπή για την Τινησία ήδη έχει προταθεί. Έτσι ώστε όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να δώσουμε όσο δυνατόν ισχυρότερη αλλά και καταλληλότερη όθηση σε όλα αυτά. Να δοθεί δηλαδή το μήνυμα ότι η, το κύριο ενδιαφέρον, η κύρια δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι χώρες αυτές είναι η οικονομική τους κατάσταση. Γι' αυτό εδώ προς στιγμή πολλοί νέοι πολιτικοί παράγοντες και κόμματα αντιμετωπίζουν πολύ δύσκολη κατάσταση και πρόβλημα. Παραδείγματος χάρη στην Αίγυπτο και την Ισία ο τουρισμός ήταν μέχρι τώρα η κύρια ο κύριος πόρος, αλλά έχασαν μεταξύ 30 και 50% του πόρου αυτού. Και από ό,τι βλέπουμε δεν μπορέσαμε να πείσουμε τους τουρίστες να επανέλθουν στις χώρες αυτές. Σε αυτήν την ειδική επιτροπή λοιπόν η Task Force πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια οι επενδυτές, οι δημόσιες τράπεζες όπως η ΕΤΕ και άλλες να πιστούν να επενδύσουν εκεί. Τρίτον, μια τρίτη παρατήρηση και τελευταία. Ποιες κατευθυντήριες γραμμές θα μπορούσαν να καθοδηγήσουν την προσπάθειά μας. Τι στάση δηλαδή γενικότερα πρέπει να τηρήσουμε προς τις χώρες αυτές που έχουν τόσες διαφορές. Πρέπει να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Τα πολιτικά πράγματα εκεί είναι τελείως καινούρια. Εμείς συνήθως τα βλέπουμε λίγο γελιογραφικά το Ισλάμ κατά της δημοκρατίας. Πολύ συζητιέται αυτό. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει κάτι ευρύτερο που πρέπει να κατανοήσουμε. Πρόκειται για μια νέα γενιά πολιτών που αρχίζει την πολιτική της ζωή με τελείως καινούριο πνεύμα και νοοτροπία σε σχέση με τους προκατόχους της. Είναι τα παιδιά του Ιντερνετ και πολλές φορές είναι πολύ έξυπνοι άνθρωποι και στην Ισία και στην Ευρώπη και αναρωτιούνται ακόμα πού θα πάνε τα πράγματα και πού θα τους οδηγήσουν τα κόμματα. Υπάρχουν εκεί δηλαδή ανθρώπινοι πόροι που μπορεί και να μην χρησιμοποιηθούν όσο θα έπρεπε από τα κόμματα. Μέσα στην μουσουλμανική αδελφότητα αναρωτιούνται αν θα χρειαστεί να ζητήσουν από όλα τα πολιτικά κόμματα να ακολουθούν το Κοράνι ή αν θα ανοίξουν το κόμμα τους και σε άλλες ιδέες που μπορεί να μην είναι ακριβώς οι ίδιες με, τον... με τις δικές τους. Αυτή η νέα γενιά λοιπόν πολιτών θα δούμε αν θα ακολουθήσει την πολιτική του ενός ή του άλλου. Ε, αυτό φαίνεται όταν συνομιλεί κανείς με νέους από την πλατεία Ταχρήρη, με νέους την Ίσιους, ότι αυτό αναρωτιούνται. Πίσω από αυτά που φαίνονται λοιπόν, εγώ είμαι στο 3-2 τώρα λοιπόν, υπάρχει το θέμα του πώς θα δημιουργηθεί ένα ολόκληρο καινούριο μοντέρνο σύγχρονο κράτος που να διαχειριστεί όσο το δυνατόν καλύτερα την καινούργια οικονομία. Τεράστια λοιπόν τα προβλήματα είναι πώς θα οικοδομηθεί μια σύγχρονη δημοκρατία, ένα σύγχρονο κράτος αν η αντιμετώπιση θα είναι πιο κοσμική ή όχι και όπως είπε και ο Επίτροπος Φίλε και για τα λίγο εδώ, εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε, να μιλήσουμε με αυτούς τους ανθρώπους με ανοιχτό μυαλό, αλλά παρακολουθώντας ταυτόχρονα στενά τι γίνεται εκεί, για να καταλάβουμε το νόημα αυτών των αλλαγών που είναι κάτι το τελείως καινούριο σε σύγκριση με το παρελθόν. Ίσως μακρηγόρησα, ζητώ συγγνώμη και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Δημό. Δώδεκα έχουν στήσει το λόγο. Θα σας παρακαλέσω να παραμείνετε στα χρονικά όρια που είχαμε και σήμερα το πρωί, δηλαδή δύο λεπτά. Ο κύριος Γκέμπς από τη Βουλή των Κοινοτήτων σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια ερώτηση έχω. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε πώς ε, το έργο μας στην υπηρεσία εξωτερικής ε, δράσης θα είναι συντονισμένο με τη δουλειά που κάνουν ε, οι εθνικές κυβερνήσεις. Σας ευχαριστώ για αυτήν την εξαιρετική ερώτηση. Η κυρία Ντεκάιζερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε όσο ο κύριος Φίλε όσο ο κύριος Βιλμό μας υπενθύμησαν πως ο οικονομικός άξονας είναι πολύ σημαντικός για να μπορέσουμε να αναγνώσουμε τις ε, αραβικές επαναστάσεις και αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε για την οικονομική τους ανάπτυξη είναι η προσπάθεια να απομακρύνουμε τους ε, πιο ε, ακραίους ριζοσπαστικούς Ισλαμιστές διότι ε, η ακραία φτώχεια είναι αυτή που επέτρεψε στα κινήματα αυτά να υπάρξουν. Η κοινωνία εκεί έχει μεγάλες δυνατότητες προσαρμογής. Ε, σκέφτομαι την ε, Παλαιστίνη, διότι τη στιγμή που άνοιξαν τις, τους εκλογικούς καταλόγους, γεγονός ότι δέχθηκαν κάποια ισλαμικά κόμματα χριστιανούς, διότι ήθελαν να φτιάξουν έναν παρόμοιο συνασπισμό. Μία ερώτηση του κύριο Φίλε. Ε, μεταβήκατε στο Μαρόκο. Μας ε, φέρατε ειδήσει καλές και λιγότερο καλές ε, και το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο είχε αρνηθεί την Συμφωνία Αλίας. Να σας ζητήσω λοιπόν πώς έγινε αντιληπτό κάτι τέτοιο, τι συνέχεια δίνεται και Εάν ε, μπορείτε να εξηγήσετε, να ανοίξετε τη συζήτηση για το ζήτημα της Δυτικής Σαχάρας ε, που βρίσκεται πίσω από τους λόγους άρνησης αυτής της ελευτικής συμφωνίας. Και δεύτερον, προς τον κύριο Βημό, δεν ακούσαμε τίποτα για τη Συρία σήμερα. Υπάρχουν νέες οικονομικές κυρώσεις ε, της Ευρώπης, αλλά υπάρχει και μια παραφωνία ε, απαράδεκτη, ε, ενώ το αραβικό πρόγραμμα το αρνήθηκαν, ε, λέγεται να πραγματοποιηθούν στρέμματα του Κατάρ. Η Μόσχα υπέγραψε μια συμφωνία με τη Δαμασκό για την αγορά 36 αεροσκαφών πολεμικής αεροπορίας. Ποια είναι η θέση και η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα αυτά, διότι προς μην δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ντεκάιζερ, επόμενος αγορητής, κυρία Νταλάρα. Ναι. Πολύ. Ε, η Ευρώπη, σύμφωνα με αυτά που είπατε και ακούσαμε και νωρίτερα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να είναι παρούσα την επόμενη μέρα. Ε, το λέγαμε European Neighborhood Funding, τώρα το καλούμε European Endowment for Democracy. Όπως και να το πούμε, νομίζω ότι έχει σημασία να αντιληφθούμε όλοι ότι για να θύσει η δημοκρατία και να στεριώσουν αυτές οι αλλαγές απαιτείται ανάπτυξη και κοινωνικό μέρισμα που θα διαχειθεί στους λαούς των χωρών αυτών. Δεν μιλάμε απλά για οικονομική ευρωπαϊκή βοήθεια. Κατά την άποψή μου μιλάμε για μια τεράστια επένδυση που θα κάνει η Ευρώπη στη νότια γειτονιά με γνώμονα τελικά το δικό μας μακροπρόθεσμο συμφέρον. Εδώ καλούμαστε να παίξουμε ρόλο και ως Εθνικά Κοινοβούλια και ως ε, ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θέλω να πω αυτό που ανέφερα ε, και νωρίς κύριε Επίτροπε στον κύριο Λεόν ότι έχει τεράστια σημασία και σας ευχαριστούμε που, που ενισχύετε την παρουσία μας εδώ. Είπατε πριν, κύριε Επίτροπε, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μεγάλη ευθύνη για τη σταθερότητα στην περιοχή και αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Γι' αυτό στην στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών η Ευρωπαϊκή Διπλωματία οφείλει να διασφαλίσει ότι αντί συγκρούσεων θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας αυτό είναι εφικτό, δεν θα κάνουμε ταμείο τώρα, δεν θα επενδύσει κάθε χώρα. Σημασία έχει η ειρήνη και η εδραίωση της δημοκρατίας στην περιοχή. Ευχαριστώ. Thank you, Mrs. Dallara. Ευχαριστούμε κυρία Δαράρα. Thank you so much, Mr. President. I'd like to ask uh, Commissioner Fula. Uh, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο φίλε, μια που σας ρώτησε και η κυρία Ντεκάιζερ για το Μαρόκο και τη Δυτική Σαχάρα, σήμερα στην Επιτροπή Εξωτερικών ε, εγκρίναμε την έκθεση για ένα καθεστώς ε, εγκύτερη συνεργασίας με το Μαρόκο. Και αυτό το θεωρούμε ως μια ευθύνη και για τις δύο πλευρές και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να πείτε κάτι για την Δυτική Σαχάρα όσον αφορά τι συνέπειες που θα έχει στην περιφερειακή συνεργασία Μαρόκο-Αλγερίας και την ευρύτερη περιοχή, την Ισία και Λιβύη. Όσον αφορά τις ε, παρατηρήσεις εκλογών, θα ήθελα να σας ε, ρωτήσω εάν γίνονται αποδεκτά τα ε, γνωστά κριτήρια και αν θα γίνει αυτό και στην Τινησία. Στον κύριο Πιμόλ. Πράγματι είναι σημαντικότερο αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε ενωμένοι ως Ευρωπαίοι και όχι με εθνικό πρόγραμμα καθένας. Γι' αυτό απόρρισα για το ότι κανείς δεν τοποθετήθηκε δημόσια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίσκεψη του Προέδρου Μπασίρ στην Λιβύη. Αναρωτιέμαι λοιπόν εάν μεταφέρατε έστω και ιδιωτικά ένα μήνυμα για τις διεθνείς υποχρεώσεις της ε, Λιβύης ε, για την ε, δικαιοσύνη. Γιατί βεβαίως αυτό έχει σημασία και ο Σαΐφ Αλισλάμ έχει κατηγορηθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Όσον αφορά το Μπαχρέιν, η αντιμετώπιση μας είναι κάπως αντιφατική. Και επίσης για την Ιεμένη, τι γίνεται με τις προοπτικές απομάκρυνσης του Αλσαλέχ. Ε, ε, ευχαριστώ κυρία Γκόμες, ο κύριος Ντόρκαμ από την Ιρλανδία. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να συγχαρώ τους μιλητές μας, ε, τόσο για σήμερα το πρωί όσο και για την την συνεδρία. Θα δούμε τα φώτα από μια διαφορετική οπτική γωνία. Πολλοί θεωρούν ότι η Αραβική Άνοιξη αποτελεί απειλή. Εγώ τη βλέπω ως πρόκληση ειδικά αυτήν την ε, περίοδο όπου αυτό λοιπόν είναι ένα, μια δοκιμασία και να δούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση τι μπορεί να πράξει προκειμένου να βοηθήσει τις χώρες αυτές χωρίς ε, επέμβαση στα εσωτερικά τους και χρησιμοποιώντας ε, τις πιο τέλειες τεχνικές της διπλωματίας να παρουσιαστεί η Ένωση μέσω των στόχων της πολιτικής γειτονία με έναν τρόπο θετικό και έναν τρόπο που δεν θα απειλεί. Αυτό λοιπόν θα είναι το σημαντικότερο κληροδότημα το οποίο μας δίνει η εποχή αυτή. Πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι για η δημοκρατία για έναν μπορεί να είναι τυραννία για άλλον. Θα πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε πως μετά από τις εξελίξεις της χώρες, πάντα θα υπάρχουν απογοητευμένοι, πάντα θα υπάρχουν ε, πρόσωπα τα οποία προσπαθούν να δημιουργήσουν ε, αστάθεια. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να το έχουμε συνεχώς κατά νου και να διασφαλίσουμε πως ε, οτιδήποτε μπορούμε να πράξουμε ως Ένωση θα πρέπει να το πράξουμε ομού, από κοινού. Είναι τεραστίας σημασίας η Ευρώπη να δρά ως ένα πρόσωπο Μόνο έτσι λοιπόν θα δώσουμε μια πολύ θετική εικόνα στην κράτη αυτά. Ευχαριστώ κύριε Τάκα, κύριο Λάμπστορφ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω με τον τελευταίο μιλητή από την Ιρλανδία. Έχω δύο ερωτήσει. Το ένα προς τον κύριο Βήμο, το... η δεύτερη ερώτηση προς τον ε, κύριο Φίλε. Προς τον κύριο Βήμο, ήσασταν πρέσβη στην Ουάσιγκτον πριν γίνετε Γενικός Γραμματέας της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικών Υποθέσεων, πρέσβης της Γαλλικής Δημοκρατίας. Στα ταξίδια σας τώρα στην Βόρεια Αφρική αντιλαμβάνεστε μια διαφορετική ματιά στην Ευρώπη όχι προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προς την Ευρώπη. Όσον αφορά, παραδείγματο χάρη, τον πρόεδρο Σαρκοζή, ο οποίο ήταν κινητήριο δύναμη πριν, ε, πίσω από την αλλαγή καθεστώτο στην ε, Λίβη μαζί με τους Βρετανού, ενώ οι θελημένα οι Αμερικανοί έπαιξαν πολύ συγκρατημένο ρόλο. Βλέπετε λοιπόν μια νέα αντιμετώπιση τη ε, Ευρώπης στη Μεσόγειο ανάλογη με τον ρόλο της στα Βαλκάνια. Ε, τώρα προς τον ε, κύριο Φίλε θα σας μιλήσω αγγλικά γιατί ε, θέλω να πω ακριβώς αυτό το οποίο είπατε στο τέλος της παρέμβασής σας. Μιλήσατε για μοναδική διπλωματική λεπτεστησία, είπατε, ελπίζετε πώς θα ξεκινήσει να βρίσκει έργα κτλ. κτλ. Ε, τι θα γίνει, πώς θα, πώς, θα, πώς θα το κλείσουμε αυτό το μαγαζάκι επιτέλους. Το Εσείς κάνετε τη δουλειά σας, ο Πιέρ Βιμόν κάνει τη δουλειά του. Αυτή η υπόθεση δεν ξέρω τι σκοπεύει να κάνει. Δηλαδή, άμα ψάχνουμε ακόμα τα έργα για να ξεκινήσει να δουλεύει, τι κάνουμε. Σας ευχαριστώ, κύριε Λάμσδορφ, νεοφύτου. Ο κύριος Νεοφύτου από την Κύπρο. Ευχαριστώ. Ο Επίτροπος κύριος Φούλε μίλησε ότι από εδώ και μπρος η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα επιδεικνύει ανοχή σε μη δημοκρατικά καθεστώτα. Και πρέπει να δείχνουμε μια απόλυτη, ένα απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Φυσικά πρέπει να κάνουμε και την αυτοκριτική μας, γιατί εδώ και δεκαετίες είχαμε συνεργασίες με μη δημοκρατικά καθεστώτα. Αλλά και αυτή η θέση, για να είναι αξιόπιστη, πρέπει να ακολουθούμε μια ενιαία πολιτική. Δεν είναι αρκετό να λέμε ότι στην Αίγυπτο, στην Τινησία, άσταση στον Μπαχρέιν, η οποία πνίγηκε στο αίμα. Πρέπει να τη σχολιάσουμε και αυτή. Και ποια θα είναι η θέση μας για χώρες όπως η Σαουδική το Κουβέιτ. Και αυτά είναι δικτατορικά καθεστώτα. Και κάτι τελευταίο είναι ε, αναφερθήκατε για το 89 και τις επαναστάσεις στον πρώην Ανατολικών Μπλοκ. Αυτές οι επαναστάσεις όμως σήμερα διαφέρουν πολύ. Εδώ δεν διασφαλίζεται η δημοκρατία μόνο με την δημοκρατικές διαδικασίες εκλογής. Οι δίκαιες και αδιάβλητες εκλογές δεν διασφαλίζουν τη δημοκρατία σε αυτές τις χώρες. Και υπάρχει ορατός ο κίνδυνος οι δημοκρατικές αρχαιρεσίες να είναι το όχημα όπου ο Ισλαμισμός θα είναι το τέλος της πράξης όπως είχαμε το παράδειγμα στο Ιράν με την πτώση του Σάχη και τις δημοκρατικές διαδικασίες που ακολούθησαν. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ε, Ευχαριστώ κύριε Νεοφίτου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι φίλοι μας από τα Εθνικά Κοινοβούλια τόνισαν την ανάγκη της συνεργασίας μέσα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών θεσμών και φυσικά και σε επίπεδο εθνικών κυβερνήσεων. Θέλω όμως να το επεκτείνω κάπως αυτή την έννοια της συνεργασίας γιατί τα καθήκοντα, τα προβλήματα της Αραβικής Επανάστασης είναι τόσο μεγάλα που καμία χώρα δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει από μόνη της. Ερωτώ λοιπόν συγκεκριμένα για μια χώρα που η επιρροή της στην περιοχή αυξάνεται συνεχώς μέρα με τη μέρα, η, του, την Τουρκία. Προσπαθούμε να την πλησιάσουμε στην Ένωση διότι ακολουθεί ήδη το δρόμο της διεύρυνσης. Ερωτώ λοιπόν πώς μπορούμε να συνεργαστούμε συγκεκριμένα, εάν πρέπει να συνεργαστούμε με την Τουρκία. Η Τουρκία για τις περισσότερες χώρες μέλη του Αραβικού Συνδέσμου είναι πρότυπο γιατί σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα πολιτικά δικαιώματα, είναι πιο δημοκρατική από τις αραβικές χώρες, υπάρχει περισσότερη ένωμη τάξη και καλύτερη οικονομία, που είναι ακριβώς η στόχη της Αραβικής Επανάστασης, περισσότερα ανθρώπινα δικαιώματα, περισσότερη δημοκρατία, πιο αποτελεσματική διακυβέρνηση και βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και του βιωτικού επίπεδου. Ο κύριος Βημών ανέφερε την Τινησία, ανέφερε την Αίγυπτο και ότι έχασαν πολλούς από τους τουριστικούς των πόρους. 50 δισεκατομμύρια πριν την ε, πανάσταση, την Ισία και τώρα τα μισά. Μέχρι το καλοκαίρι, η Αίγυπτος, μέχρι το καλοκαίρι μπορεί να χρεοκοπήσει δηλαδή. Ερωτώ, τι θα κάνουμε για να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές να ανακτήσουν μια πιο αποτελεσματική οικονομία. Φυσικά μπορούμε να κάνουμε περισσότερες επενδύσεις για εμπορικές ανταλλαγές. Να μου πείτε. Ευχαριστούμε κύριο Κόφωτ. Ευχαριστώ και εγώ για τις παρουσιάσεις αυτές. Συμφωνώ ότι πρέπει να δώσουμε πολύ περισσότερη βοήθεια στην κοινωνία των πολιτών και η πολιτική γειτονία μας για την οποία μιλούμε πολύ να παραμεταφραστεί περισσότερο σε πράξη και για την ίδια την Ένωση και μέσα στα κράτη της. Πρόκειται βέβαια για μακροπρόθεσμη προσπάθεια η στήριξη δηλαδή μιας ανεπτυγμένης πολιτικής και οικονομικής κουλτούρας Πρέπει να δημιουργηθούν οι πολιτικές δυνάμεις που θα δημιουργήσουν αυτόν τον στόχο. Χρειάζεται ανάπτυξη και από την πλευρά της Ένωσης πρέπει να το πάρουμε αυτό πολύ σοβαρά. Αν δεν μπορέσουμε να στηρίξουμε τις μεταρρυθμίσεις σε χώρες όπως η Αίγυπτος, και αν συνεχίσουν εκεί οι στρατιωτικοί να ελέγχουν την οικονομία δεν θα λυθεί το πρόβλημα του τουρισμού και θα απογοητευτεί πολύ ο λαός της αλλά και εμείς γιατί τα δημοκρατικά μας ιδεώδη θα έχουν πέσει στα σκουπίδια άμα είναι έτσι. Πρέπει λοιπόν να έχουμε να δώσουμε μία βοήθεια στις προσπάθειες αυτές, αλλά επίσης να διασφαλιστούν και να στηριχθούν οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται, ώστε τα οικονομικά συστήματα χωρών όπως η Αίγυπτος με τον τεράστιο ρόλο των στρατιωτικών να μεταρρυθμιστούν και να μπορέσει να αναθερμανθεί η οικονομία της χώρας. Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε το άνοιγμα των αγορών και άρα να στηρίξουμε όλες τις αλλαγές που θα ωφελήσουν τον λαό. Η, Ευρώπη, η Αίγυπτος αντιμετωπίζει δύσκολη κατάσταση αλλά είναι κατορθωτή η αναθέρμανση της οικονομίας της. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Γενική Γραμματέα, παρουσιάσατε πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν με τα μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Δυστυχώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Αν δείτε το τι έχουμε να κάνουμε στο εσωτερικό και το τι γίνεται, δεν νομίζω πως ε, μπορούμε να αποτελέσουμε και πρότυπο για τις ε, νέες αυτές χώρες. Η ΔΕ είπα είναι σε προεκλογική εκστρατεία και αν δείτε τους υποψήφιους των ε, Ρεπουμπλικανών δεν, ξέρετε, δεν ξέρει κανείς αν είναι κομμωδία αυτό το οποίο παρακολουθούμε ή αν είναι σοβαρά αυτά τα επιχειρήματα τα οποία λένε τώρα όσον αφορά την Τινησία και την Αίγυπτο. Συνοψίζοντας, ψωμί θένει άνθρωποι, δηλαδή δουλειά, ε, βραχυπρόθεσμα, αλλά και μεσοπρόθεσμα το τι θα γίνει να δούμε με αυτές τις χώρες. Όσον αφορά τώρα το που θα καταλήξουν οι εκλογές της ε, Αιγύπτου. Είναι πάρα πολύ νωρίς να κρίνουμε, αλλά οπωσδήποτε αυτοί οι οποίοι ξεκίνησαν αυτή την ε, διαδικασία, οπωσδήποτε δεν ε, είχαν κατά νου επιστροφή στο Μεσαίωνα και ριζοσπαστικές ισλαμιστικές δομές. Τι μέσα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν για να εργαστεί ειδικά με την νεολαία για να μπορέσει να βοηθήσει να οικοδομηθούν αυτά τα κράτη και να μην περάσουμε σε μια παλιά απικιακή, εάν θέλετε, μανιέρα και τρόπο λειτουργίας, αλλά ένα νέο τρόπο σκέψης. Αυτά και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Κράισλ Ντέρφλερ. Κυρία Φλότρο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πιστεύω πως φυσικά θα πρέπει να απευθύνουμε τις ερωτήσεις ε, για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, αλλά βλέπω να υπάρχει μια παγίδα εδώ, την οποία μπορούμε να πέσουμε όλοι. Θα ήταν παράδοξο να, πάρουμε, να ασχοληθούμε με το θέμα της θυνησίας, όπου πολλές, για πολύ καιρό ξεχάσαμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, αναφέροντας ότι η Τινησία αποτελούσε ένα οικονομικό θαύμα. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να μην βρούμε ένα νέο τρόπο και λόγο να θέσουμε σε δεύτερη μοίρα τα ζητήματα του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο όνομα της ανεργίας, της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Αυτό που μας λένε αυτές οι επαναστάσεις είναι ότι τα δικαιώματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους είναι αδιέρετα και είναι οικουμενικά. Λοιπόν, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μην ξεχάσουμε ποτέ αυτό το στοιχείο, διότι θα είναι απίστευτο το οικονομικό θαύμα της θυσίας να καταδείξει σε οικονομικό μαρασμό και να ε, ε, δοθεί ευκαιρία να μπουν στη δεύτερη μοίρα αυτά τα ζητήματα. Επειδή συζήτησα το ζητήματα θα σε βάθος με όλους ε, με όλα τα μέλη της αντιπροσωπείας μας στην Την ε, είδα ότι δεν είναι εύκολο και να υλοποιηθούν και δεν είμαι σίγουρη ότι μπορούμε να οργανωθούμε κατάλληλα προκειμένου να ε, πετύχουμε τους στόχους μας. Ε, ένα παράδειγμα να αναφέρω. Σήμερα στην Ισία έχουμε την συντακτική συνέλευση ε, η οποία απαιτεί μια διάρθρωση και επαφή με την κοινωνία των πολιτών. Μια κυβέρνηση η οποία θα εφαρμόσει νέες νομοθεσίες για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, των αστυνομικών δυνάμεων, του τύπου και ούτω καθεξής. Αυτό που θα ήταν χρήσιμο σε Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να μπορέσουμε να στηρίξουμε την σφαιρική στρατηγική, δηλαδή την νομοθετική διαδικασία, τους μηχανισμούς εμπλοκής της κοινωνίας των πολιτών, την στήριξη της κοινωνίας των πολιτών και τα ε, συνταγματικά στοιχεία. Και εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση τότε θα δράσουμε αποτελεσματικά. Θα έχει έννοια και νόημα η ε, ε, παρέμβασή μας σήμερα στην Τινησία η ομάδα μας έχει χρησιμοποιήσει σημαντικά ποσά, σημαντικά μέσα, εργαλεία, στήριξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χρηματοδοτήσει κλπ. Και κάθε ένας ε, από τους υπαλλήλου ασχολείται με τα δικά του δήματα, με τα δικά του προγράμματα, σχέδια κλπ. Πρέπει να βοηθήσουμε αυτές τις, αυτούς τους ανθρώπους, πρέπει να δουλέψουν ομαδικά, να καθορίσουμε τρεις ή τέσσερις κατηδίνες γραμμές δράσει γύρω από τι οποίε το σύνολο των προγραμμάτων και των δράσεων θα ε, μπορέσουν να προωθηθούν. Δεν ε, θα πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί με μια χώρα ή λιγότερο αυστηροί από ότι με μια δημοκρατία. Δεν πρέπει λοιπόν να κάνουμε τα σφάλματα του παρελθόντος. Ε, λοιπόν, τονίζω, υπάρχει κάτι το καινούριο που θα πρέπει να εφεύρουμε, αλλά εν πάση δεν ε, θέλω να σας κάνω κανένα μάθημα εδώ, απλά τα αυτά τα οποία λέω είναι τεχνικής συστήματα. Πρέπει επί να έχουμε ομάδες που θα έχουν τα απαραίτητα μέσα για να λειτουργήσουν διαφορετικά και φυσικά περισσότερα πρόσωπα διότι στην Ισία πραγματικά τους έχει ξεπεράσει το, η κατάσταση. Θεωρώ λοιπόν ότι ανάμεσα στην υπηρεσία εξωτερική δράση και τι υπηρεσίε τη Κομισιόν θα πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλος συντονισμός γύρω από κρατικές στρατηγικές γραμμές για να είμαστε αποτελεσματικοί. Αυτό είναι το ζήτημα. Ευχαριστώ κυρία Φλότρου. Παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο εργασία, ε, ομιλία συγγνώμη, διότι δυστυχώς ο κύριος Βιλμό θα πρέπει στις 16.30 να αποχωρήσει. Πρέπει λοιπόν στις 4.20 να ολοκληρώσουμε τις ε, ερωτήσεις για να μπορέσει να απαντήσει. Έχουμε ακόμα άλλα τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά άτομα. Ο κύριος Νταλμάνι από την Βουλή του Βελγίου. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας στην ωραία αίθουσα. Έχω τρεις μικρές ε, σύντομες μάλλον ερωτήσεις. Ε, πιστεύω ότι ο μεγάλος φόβος σήμερα στην Ευρώπη είναι η άνοιξη των ελευθεριών να μην, είναι σε, να μην μετατραπεί σε χειμώνα ε, δικαι, δικαιοκτόνο ή δικαιωματοκτόνο. Ε, ακούσαμε διάφορες απόψεις και Παράλληλα με την οικονομική συνεργασία θα πρέπει να υπάρξει ένας ισχυρός πολιτικός διάλογος. Δεν θα πρέπει να ζητάτε να ε, ε, βάλουμε πλάτη για την οικοδόμηση της δημοκρατίας και σήμερα να μας ε, ζητάτε να κλείνουμε τα μάτια σε θέματα ελευθερίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας. Νομίζω ότι αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία στον διάλογο που θέλουμε να δημιουργήσουμε, τώρα είτε πρόκειται για οικονομικά προγράμματα, είτε προγράμματα τη κοινωνία των πολιτών, θα πρέπει να δημιουργήσουμε ε, συσχετισμού, συνδέσμους ε, στο ε, οικονομικό επίπεδο. Έχουμε κοινά συμφέροντα, θέματα περιβάλλοντο, ενέργεια, γεωργία. Θα πρέπει λοιπόν να προωθήσουμε μεγάλα ενεργειακά προγράμματα στη Λεκάνη και το ίδιο σε θέματα κοινωνία των πολιτών. Θα πρέπει να αναμειχθούν αυτέ οι κοινωνίε των πολιτών. Θα πρέπει οργανώσει δικέ μα όποιος και αν είναι, αθλητικοί σύνδεσμοι, πολιτιστικοί σύνδεσμοι κλπ. θα πρέπει να αποκτήσουν σχέσεις με τους ε, αντιστοίχους ε, στις χώρες αυτές. Θα πρέπει λοιπόν να κυκλοφορούν τα πρόσωπα μεταξύ Ευρώπης και της ε, Βορείου Αφρικής. Πιστεύω ότι πολλές γυναίκες βρισκόντουσαν στους δρόμους και στις πλατείες δεν θα πρέπει τώρα να τις αφήσουμε να μπουν στη δεύτερη μία. Θα πρέπει να υπάρξουν ειδικά προγράμματα για αυτές τις γυναίκες, για είναι γυναίκες γενικότερα τώρα, για το εκλογικό ζήτημα. Ε, παρακολουθώ τις ε, αποστολέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Κομισιόν συγκεκριμένα, το γεγονό είναι ότι δεν συνάγουμε πάντα τα απαραίτητα πολιτικά διδάγματα. Ε, π.χ. Κονγκό. Έγινε εξαιρετική εργασία, αλλά κανένα πολιτικό συμπέρασμα. Θα πρέπει λοιπόν να μπορούμε να συναγάγουμε κάποια συμπεράσματα και κάποια διδάγματα. Ευχαριστώ κύριε Νταλμάνι. Είμαι υποχρεωμένος να περιορίσω το χρόνο μιλία σε 1,5 λεπτό για τους υπόλοιπους. Διαφορετικά δεν θα έχουμε χρόνο να ακούσουμε τις απαντήσεις ε, του κυρίου Βιλμό. Κυρία Μπράνερ. Ε, ναι. Ευχαριστώ Και εμένα με ενοχλεί ότι μιλάμε πάλι μόνο για απειλέ. Είναι ένα σημάδι ότι πρέπει να δουλέψουμε σκληρότερα. Πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο, να είμαστε καλύτεροι και πιο αποτελεσματικοί. Και επί τη ευκαιρία για το τελευταίο σχόλιο που κάνετε για την ευρωπαϊκή αξία, τι ευρωπαϊκέ αξίε. Εδώ μιλάμε για οικουμενικέ αξίε στην διακήρυξη των Εθνών. Εάν ε, μας, ε, πούμε ότι ε, σα φέρνουν τι ευρωπαϊκές <laughs> αξίες θα μα κλείσουν την πόρτα Αμέσω μόνο για οικουμενικέ αξίε, παγκόσμιες αξίε θα πρέπει να μιλήσουμε και να τη στηρίξουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία. ένα σύντομο σχόλιο όσον αφορά τα νέα μέσα αυτά. Αρκετά καλά, αλλά εγώ δεν βλέπω κάποια επανεξέταση των παλαιών κονδυλίων που είχαν προγραμματιστεί. Δεν έχουμε νέα ενδεικτικά προγράμματα, τα σχέδια δράσης ε, κινούνται αργά, δεν βλέπω κάποια αλλαγή σε Αλγερία, Ιορδανία κτλ. Και πρέπει εδώ πέρα να είμαστε επικριτικοί. Όσον αφορά την Αίγυπτο, επίσης ε, για το ΣΚΑΦ ε, θα πρέπει να είμαστε πιο επικριτικοί. Γιατί, αν, γιατί θα πούμε και για τους ολαυστές και τα λοιπά. Εάν δεν πούμε κάτι τώρα δεν θα είμαστε αξιόπιστοι στο μέλλον. Και με ενόχλησε το ότι είδα την ενημέρωση ε, τύπου του επικεφαλής της αντιπροσωπείας στην Αίγυπτο που έλεγε είναι επανάσταση, ακόμα καλά είναι τα πράγματα, μην ανησυχείτε για το τι κάνει ο στρατός, σοβαρά. Εγώ σοκαρίστηκα. Δεν ναι. είναι αυτό το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να ασκήσουμε κριτική. Και εξεπλάγει... Τώρα μιλήσατε για ένα European Endowment for Democracy. Αυτά. Ευχαριστώ κύριο Μπούζεκ. Mr. Chairman, welcome to the European Parliament. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τους δύο μας ομιλητές. Ξέρω ότι η σταθερότητα πρέπει να βασίζεται στη δημοκρατία, την ευημερία και την αλληλεγγύη, αλλά έχω δύο σύντομα ερωτήματα. Αλληλεγγύη. European Union. Στα Σούσα οι πρόσφυγες ζουν σε ένα στρατόπεδο εκεί σε... Τι θα κάνουμε για να βοηθήσουμε την κατάσταση αυτή στην Τινησία με τις εκατοντάδες χιλιάδων προσφύγων που δεν μπορούν να επιστρέψουν. Θα ήταν μεγάλο, μεγάλη χειρονομία αλληλεγγύης όχι μόνο για την, προς την Τινησία αλλά για ολόκληρη την Αφρική γιατί πριν από μισή μήνε το συζήτησα με τον Βόρειο Υπουργό της Δημιουργία, γιατί πήγα εκεί σε αυτό το στρατόπεδο και δεύτερον για την δημοκρατία. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολη η οικοδόμησή της. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι Εθνικές Βουλές μαζί με την Κομισιόν πρέπει από κοινού να κάνουν επισκέψεις μελέτης στις χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πρώην πρόεδρε Μπούζε και κυρία Ρομέρο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Τρεις ερωτήσεις. Πρώτον θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Φούλε και τον κύριο Βιλμούν τι μπορεί να κάνει η Κομισιόν ώστε να βοηθήσει στην διάρθρωση της ε, αντιπολίτευσης στην ε, Συρία και πώς ε, μπορεί να σταματήσει αυτός ο φαύλος κύκλος των εξοπλισμών που προετοιμάζει τον πόλεμο. Μπορούμε λοιπόν να ενισχύσουμε την, αντιπολιτικό συμβούλιο στην ε, Συρία και, κάτι, Συρία και ακόμα. Όπως είπε η κυρία Φιλότρου, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την συνεργασία μας με την Ισία και να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς ε, τα τεκτενόμενα, να ενισχύσουμε τις ομάδες μας, διότι αυτό το μοντέλο η επικράτηση αυτού του μοντέλου είναι κάτι το οποίο θα αποτρέψει τον Ισλαμισμό που μπορεί να μετατραπεί σε θρησκευτική δικτατορία. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ενισχύσουμε τις ομάδες που βρίσκονται στην Τινησία και ε, οι οποία συμμετέχουν η Κομισιόν, το Συμβούλιο για να ενδυναμώσουμε αυτή την ε, παρουσία μας στην Ισία. Και τρίτη ερώτηση. Έχει σκεφτεί ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν, μια στρατηγική για τις χώρες του Νότου που είναι υποχρεωμένες τώρα να αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις την απελευθέρωση του εμπορίου που θα προκληθεί προκειμένου οι χώρες αυτές να αναπτυχθούν. Έχετε υπόψη μια στρατηγική για την Ισπανία, για την Ιταλία, την Ελλάδα. Για αυτές τις χώρες λοιπόν που από πλευράς ε, γεωργίας, ε, ε, μεταπητικής βιομηχανίας έχετε σκεφτεί μια στρατηγική για τις χώρες αυτές του Νότου. Η κυρία Μπενελά το λόγο. Έχουμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε ερώτησή μου απευθύνεται στον κύριο Φούλε. Μιλήσατε για την αύξηση των υποτροφιών Μον ε, Μούντι, αλλά θα πρέπει να ενημερώσετε τα κράτη-μέλη για το θέμα των ε, προξενικών θεωρήσεων. Διότι αν ε, δεν υπάρχουν αυτές οι θεωρήσεις τότε χάνουμε αξιοπιστία για την Αλγερία. Η Αλγερία είναι μια χώρα πολύ σημαντική, παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Είχα την ευκαιρία να μεταβώ στο Αλγέρι στα τέλη του Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου και δεν μπορώ να καταλάβω πώς λέτε ότι είστε ε, ικανοποιημένος που σας προσκαλούν οι αλγερινές αρχές. Γιατί, διότι όταν αυτά μετά αυτά που συνέβουν στην την Ισία, ο πρόεδρο του Μπουτεφλίκα θέλησε να αλλάξει τα πράγματα. Είπε, αμάν κάτι πρέπει να κάνω εδώ. Και πρόωθησε την ιδέα για την τροποποίηση του συντάγματο. Ε, οι διάφοροι νόμοι έφτασαν ενώπιον τη ε, ενθροσυνέλευσης, αλλά αυτή η ενθροσυνέλευση είναι η ίδια με αυτή που υπήρχε πριν. Δεν άλλαξε τίποτα αυτοί που είναι στη Βουλή θα αλλάξουν νόμους οι οποίες δεν είναι τίποτα άλλο παρά ε, νόμοι για που καταπατούν, θέλουν να καταπατήσουν μάλλον τα δικαιώματα. Αυτή η νόμη λοιπόν είναι ουσιαστική για την ε, επιβίωση κοινωνίας των πολιτών. Όταν πήγα στο Αλγέρι ε, συνάντησα πολλούς προσώπους της κοινωνίας των πολιτών και δεν είναι διόλου πεπισμένοι ότι υπάρχει πραγματική βούληση για αλλαγή στην χώρα. Ακούμε λοιπόν ωραία λόγια από τους βουλευτές, οι οποίοι όμως είναι οι πρώην, οι παλιοί βουλευτές, που ζητούν και δηλώνουν ότι θα κάνουν αλλαγές. Λοιπόν, το Φεβρουάριο έμαθα ότι θα στο Αλγέρι, παρακαλώ να συναντήσετε την κοινωνία των πολιτών και να του ε, ακούσετε είναι τα ευήκονου, Τι αγγείες λοιπόν εγγύες δίνεται, πω θα υπάρξει μια πραγματική δημοκρατική εκλογική διαδικασία κάτω από αυτές τι συνθήκες. Και να πω κάτι ακόμα, το 2012 είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για την Αλγερία, είναι η πεντηκοστή η τη ανεξαρτησία και ο πρώτος ε, πρωθυπουργό του Μπερθάντα Βάς έγραψε ένα βιβλίο που λέει για την κατασχεμένη ανεξαρτησία. Υπήρξε ε, όντως ε, αυτή η κατάσχεση, είναι, σωστό. Ευχαριστώ κύριε Μπαρ Ατού. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως ε, και όλοι οι ειδήσει προτιμά να υπάρξει ένα αίτημα, μια αντιμετώπιση ευρύτερη των αιτημάτων των χωρών αυτών σε πολλά επίπεδα, αλλά τελικά ε, είδαμε ότι συνεχίστηκαν οι σχέσεις με όλους τους ε, ε, όλες τις απολυταρχικές κυβερνήσεις. Εμεί θέλαμε να υπάρξει πρόοδος, αλλά το γεγονό είναι ότι και οι στους διάφορες εξεγέρσεις, στους δρόμους, πλατείες κλπ. Δεν ε, περίχαν τόσο πολύ ένα θρησκευτικό στοιχείο, αλλά τώρα βλέπουμε ότι δυστυχώς ε, τα πράγματα έχουν ξεφύγει από, από την αρχική τους ε, κατάσταση. Αυτό που με απασχολεί είναι το εξή Η Ευρωπαϊκή Ένωση να περάσει στα ψηλά τα θέματα όπως το Ισουδικής Αραβίας ή το Μπαχρέιν σαν να μην υπάρχουν. Υπάρχουν εξαιρετικέ σχέσεις όμως σε κάθε επίπεδο, πολιτικές, στρατιωτικές κλπ. Και έχουμε το παράδειγμα του Μαρόκου, το, οποίο όμως διεξήχθησαν γενικέ εκλογέ με ένα πολύ χαμηλό ποσοστό συμμετοχής, 25% συμμετοχή και ένα τμήμα της Δυτικής Σαχάρας ε, το κατέχει παρανόμως το, το Μαρόκο. Και το έχουμε σαν παράδειγμα και ρωτώ, Μάθαμε κάποιο, ε, κάποιο δίδαγμα. Ευχαριστώ. Ο κ. Κροτσέτα έχει το λόγο. Πρώτο, Κατάρ. Το Κατάρ παίζει ένα ρόλο πολύ σημαντικό και σε στρατιωτικό επίπεδο. Υποστήριξε την επέμβαση στην ε, Λιβύη, παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα μαζί με τους ε, γείτονές της, εταίρους, Σαουδική Αραβία κλπ. όπου ε, γίνονται κάθε χρόνο εκτελέσεις και γίνονται εκλογές στην Τινησία και την Αίγυπτο, το Κατάρ ε, χρηματοδοτεί όλα τα Ισλαμικά κινήματα. Το Κατάρ θυρίζεται από τις Ηνωμένες αλλά ταυτόχρονα συζητάει και με την Ισλαμική Τζιάρτη στο Μαρόκο και με τους Ισλαμιστές της όλης περιοχής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως θα πρέπει να κάνει αυτοκριτική, διότι την Ισιακή Επανάσταση ε, κοίταζε το ευρωπαϊκό μοντέλο, εμεί ε, πάντα του μιλούσαμε για δικαιώματα, δικαιώματα, δικαιώματα. Αυτό να καταλάβουμε ότι σε επίπεδο δικαιωμάτων ε, δεν υπάρχει μόνο η δημοκρατία, αλλά και το δικαίωμα των λαών στην τροφή. Και θεωρώ ότι σε επίπεδο οικονομικών σχέσεων και παρεμβάσεων που μπορούν να προσεγγίσουν τις χώρες αυτές αλλά και σε επίπεδο Ισλαμικών κινημάτων που είναι αρκετά μετριοπαθή μερικές φορές αυτό αποτελεί την απελπισμένη απάντηση σε θέματα που τους καίνε άμεσα. Ευχαριστώ, η κυρία Βερσία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ, ως Γαλλίδα, θέλω να πω ότι ας κάναμε την, ε, τον ισολογισμό, τον απολογισμό, συγγνώμη, της γαλλικής κυβέρνησης ένα χρόνο μετά. Να κάνουμε τον απολογισμό της ε, κατάρρευσης του τείχους ε, του Βερολίνου ένα χρόνο μετά. Λοιπόν, δεν θα πρέπει να βιαζόμαστε δεν πρέπει να προτρέχουμε διότι πολλά θα πρέπει να μας συγχωρέσουν οι χώρες αυτές. Θα πρέπει να δούμε τα πράγματα κατάματα αφήνοντας χρόνο στους άνδρες και τις γυναίκες που αγωνίστηκαν για την ελευθερία τους και βοηθώντας τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν δέχομαι να δίνουμε μαθήματα ούτε να κάνουμε ε, διάφορα αμαλγάματα, κάθε χώρα έχει τη δική της ιστορία. Και τελικά ας ε, σταματήσουμε να δημιουργούμε φόβους οι ε, Ισλαμιστές ως αν παντού οι, καθολικοί και οι προτεστάντες να ήταν ίδιοι. Ότι, ως αν να μην μπορούσαμε να ε, έχουμε ψουθύνει στις οικουμενικές μας αξίες, δηλαδή την ελευθερία επιλογής στις σκεπτικές μας ιδεών και να μην κρίνουμε τους ανθρώπους ε, ανάλογα με την σκεφτική τους ε, ένταξη και, Χρειάζεται λοιπόν να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές να οικοδομήσουν τη δημοκρατία τους, δίχως όμως να είμαστε πιο απαιτητικοί σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας από ό,τι είμαστε στο παρελθόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να βλέπουμε με ενδιαφέρον τα τεκτενόμενα, αλλά να μην ζητάμε περισσότερα από όσα γίνεται και έχουμε και ένα κομμάτι ευθύνη στην θέματα οικονομική βοήθεια. Σα ρωτώ κύριε Επίτροπε, κατά την περσινή χρονιά ανακοινώθηκαν τεράστια ποσά Ω ενίσχυση στι χώρε αυτές. Από ό,τι γνωρίζω, η πρώτη βοήθεια έφτασε στην Τινησία τουλάχιστον τον Δεκέμβριο. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια, μια καλή και αναλυτική ενημέρωση της βοήθειας που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει στα κράτη αυτά. Ευχαριστώ κυρία Βερζιά. Να δώσω το λόγο στον κύριο Βιλμό. Νομίζω πως ο Επίτροπος έχει λίγο παραπάνω χρόνο και ή δυνατόν θα προτιμούσε ο κύριος Βιλμό να μιλήσει πρώτος έτσι ώστε να μπορέσει να αποχωρήσει με τα χαράς Προέδρε θα αφήσω όλες τις δύσκολες ερωτήσεις στον κύριο Επίτροπο και έτσι θα μπορέσω να φύγω με ελαφρά πηδηματάκια. Ε, να απαντήσω τώρα στα ερωτήματα που ετέθησαν, δηλαδή πώς, μπορούμε, πώς φροντίζουμε μάλλον, να συντονίσουμε τη δράση μας με αυτήν των κρατών μελών. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή ερώτηση και θεωρώ ότι είναι και πολύ σημαντική, διότι επανειλημμένα ακούστηκε κατά πόσον θα πρέπει να ενισχύσουμε τις ομάδες μας, αν έχουμε τα μέσα κλπ θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι σε αυτές τις χώρες πολλά κράτη-μέλη αναλαμβάνουν δράσεις, βρουν, προωθούν προγράμματα και θα πρέπει πράγματι να συντονιστούμε. Προσπαθούμε να το πράξουμε, έχουμε επαφές με καθένα από τα κράτη-μέλη επιτόπου, οι οποίες μας συνεργάζονται με τα αντιπροσωπείες των κρατών μελών, όπως το κάνουμε και στην υπηρεσία εσωτερικής δράσης με τις υπηρεσίες της Κομισιόν, θα πρέπει όλοι να εργαστούμε προς την αυτή κατεύθυνση. Και αυτό με οδηγεί στο να πω και τέθη ένα ερώτημα από την κυρία Φλότρου, σχετικό ότι θα πρέπει να ορίσουμε ένα πλαίσιο, ένα πλαίσιο στρατηγικό αφενός σχετικά με το τι θέλουμε να κάνουμε τα προσεχή χρόνια και να έχουμε και ένα πρόγραμμα δράσης ε, για την ε, ε, προώθηση αυτού του προγράμματος και εδώ μπορούμε να δούμε τι κάνουν τα κράτη-μέλη από πλευράς τους Τώρα σχετικά με το θέμα της Task Force που ανέφερε ο Επίτροπος Φιούλε αλλά και είπα ότι εκπρόσωπος θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία των ιδιωτών του δημοσίου, ιδιωτικών και δημοσίων τραπεζών, κομισιών. Όλοι λοιπόν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε πράγματα. Θεωρώ ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και χρειάζεται να δουλέψουμε επ' αυτού με τρόπο συνεχή. Μου θέσατε το ερώτημα κυρία Κάιζερ για την Συρία. Αυτό που θα πρέπει να εξετάσουμε είναι πως οι αποφάσεις που έλαβε η ε, Αραβικός Σύνδεσμος την Κυριακή το βράδυ είναι πολύ σημαντικές. Ε, όπως γνωρίζετε η Υπουργική Επιτροπή συνήλθε και θεωρήσαμε ότι το μόνο πράγμα που θα συζητούσαν θα ήταν παρατείνεται ή δεν παρατείνεται η, αποστολή, η παραμονη των αποστολών πεσταλμένων. Είδατε ότι αποφασίστηκε να ε, παραταθεί, αλλά υπήρξαν διστάμενες απόψεις ότι δηλαδή πρέπει να αντικατασταθούν ε, κατά ένα τμήμα του τουλάχιστον. Και υπήρχε και κάτι ακόμα το οποίο δεν περιμέναμε, ήταν μια απόφαση θαραλέα ότι ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος, ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος παρουσίασε επιπλέον στοιχεία, τα οποία πάνε μακριά, διότι αυτό το οποίο δημιουργούν είναι αυτό που ονομάζαμε επιλογή της ιεμένης ε, θα πρέπει φυσικά να συγκρίνουμε τα πράγματα, αλλά αυτό το οποίο λένε, εάν διαβάζετε ανάμεσα στις αράδες, ότι ο κύριος Ασάρ θα πρέπει να αναθέσει ε, στους διαπραγματεύσει διαπραγματεύσεις έναν από τους αντιπροέδρους του, ότι θα πρέπει να πάμε προς μια, κυβέρνηση μετα, μεταβατική και θα πρέπει να δημιουργηθεί θέση ενό ειδικού απεσταλμένου του Αραβικού Συνδέσμου που συμμετέχει στι διαπραγματεύσει και πολύ πιο σημαντικό όλα αυτά θα πρέπει να αποστέλλονται στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ προς έγκριση και αυτό το πρόγραμμα λοιπόν να λάβει την στήριξη της παγκόσμιας κοινότητας μέσω του ΟΗΕ. Είδατε λοιπόν τις πρώτες ε, αντιδράσεις ε, των Συριακών αρχών, ένα κάθετο όχι, αλλά ε, ο Αραβικός Σύνδεσμος δεν σταματάει εκεί. Η Ρωσία έχει μια αντίδραση που δεν είναι αδιάφορη. Εδώ και τρεις εβδομάδες στο Συμβούλιο Ασφαλείας προσπαθούμε να συμφωνήσουμε επί ενός ψηφίσματος. Πρέπει λοιπόν να παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Ε, με συμπτώσει τα πράγματα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. είπατε εκπρόσωπος Κυριάστον ε, ήταν σε συνεχή επαφή με τον Γενικό Γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Ε, δουλεύουν για να δουν πώς ε, μπορούν να τους στηρίξουν στις πολιτικές προσπάθειες, προσπάθειες πολιτικής διαμεσολάβησης. Χθε στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών του Τούστικ υπόθηκε ότι θα πρέπει να στηριχθεί η Αραβική, ο Σύνδεσμος και για μια ακόμη φορά δεν πρέπει να έχουμε ψευδεστήσεις. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Μέχρι τώρα είδαμε ότι οι Συριακές αρχές δεν ήταν έτοιμες να δεχθούν το οτιδήποτε, αλλά αυτό που προσδίδει ενδιαφέρον είναι ότι εδώ και μερικές εβδομάδες βλέπαμε ότι τίποτα δεν προχωρούσε, αλλά του Συμβούλου Ασφαλεία, ο Αραβικό Σύνδεσμο, η δήλωση των Ρωσικών Αρχών, η Κίνα, η Βραζιλία και άλλοι αρχίζουν να εκδηλώνουν μια κάποια επιφύλαξη ε, απέναντι στην ε, Συριακή κυβέρνηση και επίση κάτι άλλο που με ρωτήσατε, ναι είμαστε σε επαφή φυσικά με την ε, αντιπολίτευση της Συρίας και προσπαθούμε να τους ενθαρρύνουμε προκειμένου να συνεργαστούμε στην την αυτή κατεύθυνση και να στηρίξουμε τις προσπάθειες του Αραβικού Συνδέσμου. Ο βαρομονικό κίνησης που αντιμετωπίζουμε τώρα είναι η κατάσταση να επιδεινωθεί περαιτέρω στην Συρία και να οδηγηθούμε σε ένα φίλιο πόλεμο. Και αυτό θέλουμε να αποφύγουμε, διότι εάν συμβεί κάτι τέτοιο, αυτό θα αποβεί εις βάρον όλων συμπεριλαμβανομένων του λαού της ε, χώρας. Κυρία Γκόμες, με ρωτήσατε για την επίσκεψη του Πρόεδρου Μπασίου στη Λιβύη. Ναι, ήδη γνωστοποίησαμε στις ε, προσωρινέ αρχές της Λιβύης ότι θεωρούμε πω δεν ήταν κάτι το καλό, ε, μάλλον είναι αντίθετο προς τις διεθνείς ε, συμβάσεις και συνθήκες, το είπαμε, διότι θα αναλάβουμε και ένα πιο επίσημο διάβημα, αλλά γι' αυτό επατείται η συμφωνή γνώμη όλων των κρατών μελών, αλλά εμείς ήδη το αναφέραμε στους συνομιλητές μας, διότι δεν θα έπρεπε να χάσουμε χρόνο. Ε, ρωτήσατε για την Ιεμένη και τον Μπαχρέιν, για την Ιεμένη, και επανέρχομαι σε αυτά που είπα προλίγου σχετικά με τη Συρία, υπήρξε μια εξαιρετική ε, διπλωματική διαπραγμάτευση αλλά κατορθώσαμε να συμφωνήσουν οι χώρες του κόλπου, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, πρόσωπος, ε, ειδικός πρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και παρά όλες τις δυσκολίε να κατορθώσουμε, να προχωρήσουμε ε, και να δεχθεί ο πρόεδρος Σαλέ ήταν μια πολύ σημαντική διελκυστίδα. Ξέρω ότι, δεν, ότι πολλοί δεν ε, συμφώνησαν με την ρήτρα ατιμορρησίας, ειδικά ο λαός ε, της χώρας, αλλά εάν ε, εν τέλει θέλετε να εκδιωχθεί ένας πρόεδρος, να τον απακρίνεται από την εξουσία, μερικές φορές θα πρέπει να δοθούν κάποιες παραχωρήσεις. Τα υπόθεση δεν έχει τελειώσει, θα δούμε εκ των υστέρων. Για τον Μπαχρέιν τα πράγματα είναι περίπλοκα πριγκιπικές αρχές του Μπαχρέιν προσπάθησαν με συζητήσεις ιδιαίτερα δύσκολες ε, να βρουν κάποιο άνοιγμα. Είχαν εκθέσεις για την καταπίεση στο Μπαχρέιν πολύ ενδιαφέρουσε. η κατάσταση είναι περίπλοκη, ασταθής, πρέπει να συνεχίσουμε να ενεργούμε, να διατηρήσουμε επαφές με τις γειτονικές χώρες, Σαουδική Αραβία φυσικά και άλλες χώρες του κόλπου και αυτό έχει τη σημασία του. Ερώτηση τώρα σχετικά με την Αίγυπτο και την Τουρκία. Ειδικά για να τονίσω ότι ο κίνδυνος της Αιγύπτου ήταν η αποτυχία, η χρεοκοπία. Αλλά εδώ δεν υπάρχει ε, μυστικό, όταν μιλάμε για μακροοικονομική βοήθεια, ε, ε, ξέρετε ότι εμπλέκεται το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πρότεινε την, πρότεινε την βοήθειά του στο Στρατιωτικό Συμβούλιο για λόγους που δεν καταλάβαμε, ή μόνο που αν καταλάβαμε, αλλά θέλουμε να πούμε, είπε όχι το Στρατιωτικό Συμβούλιο και ελπίζω να το επανεξετάσουν και να το δεχθούν, γιατί Μιλάμε για 3,5 δις ε, δολάρια. Δεν είναι κάτι το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να το κάνει από μόνο της. Ε, Σίγουρα ότι ο Φίλε θα σας πει περισσότερα από ό,τι εμένα, από εγώ. Ο ρόλος μας είναι γύρω από μια μακροδημοσιονομική ενίσχυση για την στήριξη που μπορεί να δοθεί αναφορικά με την προετοιμασία των εδάφους για ιδιωτικές επενδύσεις. Τώρα για την Τουρκία, επειδή με ρωτήσατε, η επιρροή της Τουρκίας είναι θεμελιώδης στην περιοχή. Είναι περίπλοκη, είναι αφιλεγόμενη θα έλεγα, παφωτεριζουσα Ε, πολλοί ηγέτες της περιοχής λένε ότι χαίρονται για τη σχέση και τη συνεργασία με την Τουρκία. Σε ιδιωτικές συζητήσεις όμως λένε πράγματα λίγο πιο ε, συγκαλυμμένα. Πάντως είναι γεγονό ότι πρέπει να συνεργαστούμε με την Τουρκία. Γνωρίζετε, ο κ. Άστον είχε προσκαλέσει τον Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων, κ. Νταβούτογλου, χθε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων για να συζητήσουμε ε, όλα τα προβλήματα της περιοχής. Εν τέλει, ε, ο Τουρκο υπέξ αποφάσισε να ε, αναβάλει για ένα μήνα την συνάντηση αυτή με τους Ευρωπαίους ε, ομολόγους του. Θα έχουμε πολλά να πούμε με τον ε, υπέξ της Τουρκίας. Ίσως ακόμα κανένα δυο να προσθέσω ερωτήσεις που μου τέθηκαν. Ναι, η επιτήρηση των εκλογών στο Κονγκό. Πράγματι, έγινε αποτελεσματικά, οι εκλογές ε, αποδείχθηκαν διαφανείς και τίμιες, αλλά το καθεστώς δεν ακολούθησε τις συστάσεις της. Δώσαμε το μήνυμα στις αρχές της δημοκρατίας του Κονγκό ότι η συνέχεια της δημοκρατικής εκλογικής διαδικασίας είναι κάτι που θα το προσέξουμε ιδιαίτερα. Συμφωνώ και εγώ ότι δεν ήταν ικανοποιητικό το γενικό αποτέλεσμα, αλλά όπως είπαν και άλλοι, όλα αυτά είναι και θέμα χρόνου. Δεν καταλήγει κανείς σε μια σύγχρονη δημοκρατία τόσο γρήγορα, μια δημοκρατία που να μοιάζει με τις δικές μας, χωρίς κάποια εκμάθηση, χωρίς κάποιο χρόνο. Δεν πρέπει να αποθαρρυνόμαστε εύκολα με τις πρώτες δυσκολίες που θα αντιμετωπίζουμε. Κύριε Λάμπσδορφ, δύο ερωτήματα θέσατε αν δεν απατώμε. Πρώτον για την Ένωση για τη Μεσόγειο και μάλλον δέχομαι αυτά που είπατε αλλά νομίζω ότι από την Ένωση για τη Μεσόγειο μπορούν να σωθούν μερικά. Η περιφερειακή διάσταση, η ιδέα ενός μεγάλου προγράμματος που να ξεπερνάει οι συγκεκριμένες χώρες και που να αφορά ολόκληρη την περιοχή για τομείς όπως το νερό, τις μεταφορές, την ενέργεια, εκεί μπορεί ίσως να γίνει κάτι. Και τρίτον, η προσπάθεια δημιουργίας εταιρικών σχέσεων δημοσίων και ιδιωτικών πριν πούμε λοιπόν ότι τελείωσε αυτή η ιστορία, θυμηθούμε ότι υπήρχε καταρχήν η διαδικασία της Βαρκελόνης, μετά η Ένωση για τη Μεσόγειο, να μην τα πετάξουμε όλα, με ό,τι μπορεί να σωθεί ας περισωθεί. Αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και τέλος, Αφήνω στον Επίτροπο Φιούλε τις επόμενες απαντήσεις. Μου θέσατε όμως μία άμεση ερώτηση ότι είμαστε και οι δύο πρώην της Ουάσιγκτον και πρέπει να ξέρουμε τις δυσκολίες που έχει η Ευρώπη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των χωρών αυτών. Η Ουάσιγκτον καταλαβαίνει τη διαφορετική αντιμετώπιση της Ευρώπης και αυτό προσπαθούμε και εμείς να το εξηγήσουμε για τη Λιβύη. Θα σημειώσατε ότι η Λέδη Άστον κράτησε τις επαφές της και με την Αφρικανική Ένωση και με τον Αραβικό Σύνδεσμο ενώ ακούγονταν τόσες πολλές επικρίσεις για τη στρατιωτική παρέμβαση που, στην οποία συμμετέσχουν μερικές χώρες μέλη. Προσπαθούμε να οικοδομήσουμε γέφυρες και με τις χώρες αυτές και τις οργανώσεις που βρίσκονται σε αυτές να δημιουργήσουμε κάποια εμπιστοσύνη μεταξύ μας για να λυθεί έτσι κάποτε και το πρόβλημα της Ιεμένης και να δούμε τι μπορεί να γίνει και για τη Συρία και την Ιεμένη. Πρόκειται εδώ για τη δημιουργία ενός πολιτικού κεφαλαίου και ακόμη πιο τελευταίο θέμα τώρα θα ήθελα να τονίσω για τις παρατηρήσεις του Προέδρου Μπούσεκ. Ναι, πήγε και εκείνο έκανε επισκέψεις στις χώρες αυτές και αυτό είχε σημαντική επίπτωση. Μας το λένε συνεχώς οι αρχές των χωρών αυτών. Αλλά τέτοιες ανταλλαγές απόψεων και διάλογοι πρέπει να συνεχιστούν για να γίνει κατανοητό τι ακριβώς είναι η δημοκρατία. Να γνωρίζετε κύριε Πρόεδρε ότι πολλές χώρες, την Ισία, Μαρόκο και αλλού, ενδιαφέρονται ιδιαίτερα από ε, την εμπειρία σας για τον εκδημοκρατισμό και της ίδιας σας της χώρας και ότι υπάρχουν ανταλλαγές ιδεών. Πρέπει λοιπόν να μην αποθαρρυνόμαστε εύκολα γιατί υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες, πληθώρα πρωτοβουλειών που γεννιούνται στις χώρες αυτές και εμείς το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε κάποια κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε γιατί πάλι μίλησα πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Βημόν για την παρουσία του μεταξύ μας και θα δώσω τώρα το λόγο στον Επίτροπο Φίλε. Σας ευχαριστώ. Και είναι γύρω στις 15 ερωτήσεις που θα ήθελα να απαντήσω λίγο πολύ. Συμφωνώ πλήρως με κάποια από αυτά τα οποία είπατε, που υπογραμμίσατε το πόσο σημαντικό είναι να απαντήσουμε το τι συμβαίνει στον Νότο με την νέα αυτή πολιτική. Εγώ θα έλεγα πως έχουμε μια νέα πολιτική. Τώρα αν είναι η τέλεια δεν είπα αυτό. Αλλά είναι μια πολιτική. Έχουμε την ε, εταιρική σχέση για τη δημοκρατία και την κοινή ευημερία πέρσι. Την υιοθετήσαμε. Υιοθετήσαμε επίση διάφορε ανακοινώσει που τι συζητήσαμε εδώ πέρα. Γίνεται πάρα πολλή δουλειά και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην νότια διάσταση και στην διάσταση αυτή της πολιτικής μας. Οπότε υπάρχει νέα πολιτική. Επίσης έχουμε ένα νέο πλαίσιο Έχουμε ένα μέσο τη Λισαβόνα. έχουμε την υπηρεσία εξωτερική δράση, τον είπα το εκπρόσωπο, την είπα το εκπρόσωπο και αντιπρόεδρο ταυτόχρονα. Έχουμε ένα μηχανισμό συντονισμού που δεν είχαμε πριν εντό τη Κομισιόν για να συντονιζόμαστε με την υπηρεσία εξωτερική δράση και του διαφορού επιτρόπους ε, ανάλογα με τον αρμοδιότητα το καθενό. π.χ. η συνεργασία για την κινητικότητα. Αυτό δεν σημαίνει πως ε, σας εγγυώμαι πως έχουμε και νέο τρόπο σκέψης, νέους ανθρώπους. Δεν μπορώ να σας εγγυηθώ κάτι τέτοιο. Και αυτή είναι μια πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Αλλά θα έλεγα πως έχουμε καταβάλει κάθε προσπάθεια να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της ε, νότιας γειτονιάς μας. Ο συντονισμός τώρα με τα κράτη-μέλη είναι ένα θέμα κρίσιμο για να μπορέσουμε να έχουμε μια πραγματικά συνεκτική πολιτική. Η συνθήκη της Λισαβόνας δημιουργεί τις συνθήκες, αλλά δεν δημιουργεί και δεν μπορεί να δημιουργήσει ένα συντονισμό 100% μεταξύ των κρατών μελών και της υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ε, επί τη ευκαιρία η ομάδα αυτή δράση είναι το πλαίσιο ακριβώς το οποίο κατά την άποψή μου μπορεί να επιφέρει ένα συντονισμό με του Ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού Οργανισμού ε, και τα κράτη-μέλη από την άλλη. Και πολλά πρέπει να γίνουν για να ε, έχουμε αποτελέσματα. Τώρα για το Μαροκό. Υπήρχε ανησυχία. Το έχω συζητήσει με τις αρχές το τι σημαίνει μία ψηφοφορία για το πρωτόκολλο περί αλληλείας. Υπήρχαν πολλές προσδοκίες για την ψηφοφορία της Συμφωνίας Γεωργίας. Υπήρχαν λοιπόν συζητήσεις, ερωτήσεις του για το τι σημαίνει. Υπήρχαν υπήρχε το ζήτημα του σε ποιο βαθμό ε, δίνουμε πραγματική σημασία σχέση με το Μάρκο. Γιατί εν τομέα της αλληλείας φαίνεται πως είναι ικανοποιημένη με το να εργαστούμε εμείς πάνω σε μια νέα έντολη η οποία όπως τόνισα θα λάμβανε υπόψη τις ανησυχίες που εξέφερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όσον αφορά τη συμφωνία της Γεωργίας την συζητήσαμε πιο λεπτομερώς μετά από τις διαβουλεύσεις που είχαμε αρκετούς βουλευτές, ειδικά στο Στρασβούργο. Και να σας πω δύο-τρία πράγματα. Πρώτον, θα σας αφήνω μια επιστολή που θα περιγράφει τα αποτελέσματα των επιφών μου με τις αρχές του Μαρόκου, γιατί βεβαίως αφορά και τις ανησυχίες που ετέθησαν στη συζήτηση αυτή. Επίσης θα προσπαθήσω να διαλύσω κάποιους μύθους που υπάρχουν όπως το ότι το Μαρόκο δεν τηρεί τους κανόνες όσον αφορά την Συμφωνία Ελευθερου που είχαμε ήδη. Δεύτερον, είμαστε έτοιμοι και συνεργαζόμαστε με κάποιους από σας ε, για να έχουμε ένα σχέδιο ψηφίσματος το οποίο θα συνοδεύσει την ε, συμφωνία αυτή γεωργικών προϊόντων και θα ψηφιστεί λίγο πολύ ταυτόχρονα. Θέλουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα αυτή να αντικατοπτρίζει τις ανησυχίες σας, δεύτερον να είναι όσο δυνατόν πιο ρεαλιστική γιατί μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα ακριβώ πριν την ψηφοφορία να δεσμευτούμε ξεκάθαρα σε κάποιες διατάξεις, σε κάποιους όρους αυτού του ψηφίσματος για να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε το Μαρόκο να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουμε. Και ξέρετε πώς θα συνεχιστεί η δουλειά το αναμένω αυτό στην ε, ψηφοφορία του Φεβρουαρίου για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε όλες τις προσπάθειες που, που έχουν γίνει. Δεν αναφέρθηκα ειδικά στη Δυτική Σαχάρα, στην ε, περιφερειακή διάσταση, αλλά παρατήρησα πως υπάρχει μια στεδιακή διαδικασία βελτίωση των σχέσεων του Μαρόκου με την Αλγερία. Και όπως ακριβώς και με τις αρχές του Μαρόκου, έτσι θα μοιραστώ και κάποια μηνύματα με τις αρχές της Αλγερίας. Δηλαδή θέλουμε να υπάρξει μια ομαλοποίηση των σχέσεων των δύο αυτών χωρών, γιατί τότε θα ανοίξει ο δρόμος για μια περιφερειακή συνεργασία στο πλαίσιο της ε, Ένωσης ε, του Μαγκρέμπ. Θα ωφελήσει τις χώρες αυτές, την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μας επιτρέψει και το ξεκινήσαμε ήδη αυτό να προετοιμαζόμαστε δηλαδή, να προετοιμάζουμε μια συγκεκριμένη ανακοίνωση για τη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός και της Ένωσης ε, του Αραβικού Μαγκρέμπ από την άλλη. Τώρα για την ε, Ένωση της ε, Μεσογείου πράγματι χρησιμοποίησα κάποια διπλωματική γλώσσα. Καμιά φορά χρειάζεται για να περιγράψει κανείς τις ε, δυσκολίες. Και καμιά φορά έχω την αίσθηση πως υπάρχει η πρόθεση να γίνει κάτι καλό με τη δικασία της Βαρκελόνης, αλλά από εκεί πέρα όλα πήγαν στραβά. παρακολουθήσαμε εμείς ε, παθητικά ως έναν βαθμό. Το ότι δεν υπήρχε πρόοδος στην ειρηνευτική δικασία στη Μέση Ανατολή και αυτό μας κόστησε σε ενέργεια. Και δεν μπορέσαμε επίσης να επιτύξουμε πως υπάρχει μια κάποια προσθέμενη αξία και ε, πάλι ε, υπάρχει η Ένωση για τη Μεσόγειο, η οποία έχει μείνει χωρίς γενικό γραμματέα. Υπάρχει όμως μια γραμματιακή συνεργασία και μια τομεακή συνεργασία η οποία δεν υπάρχει πουθενά αλλού σε οποιοδήποτε άλλο τομέα της αρμοδιότητάς μου. Οπότε, αν είναι να ακυρώσουμε όλο το το έργο αυτό της Ένωσης για την ε, Μεσόγειο θα πρέπει να έχουμε κάποιο άλλο πλαίσιο για την τομεακή αυτή συνεργασία του Βορρά και του Νότου της Μεσογείου και ταυτόχρονα μετά από μήνες και μήνες πολιτικών συζητήσεων και κλεισμένο των θυρών. Νομίζω πως ε, είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να λύσουμε το ζήτημα. Το ζήτημα του εάν είναι κυβερνητικός, διακυβερνητικός οργανισμός, εάν πρέπει να βασίζεται στην κοινοτική προσέγγιση, αν είναι κάτι ε, ανάμεσα στα δύο, ε, τι θα γίνει με τη συμπροεδρία, χώρα από το βορρά, από τον νότο, τι ρόλο θα παίξει η υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Νομίζω πως σιγά σιγά βρίσκουμε τις σωστές απαντήσεις και θα δούμε περισσότερη υπηρεσία εξωτερική δράση, περισσότερη κοινοτική προσέγγιση και νομίζω πως αυτό θα ωφελήσει την ε, Μεσογειακή Ένωση. Για τη συνεργασία τώρα με την Τουρκία. Πολλά ακούστηκαν ήδη. Το πρόβλημα που έχουμε είναι όχι πως ε, δεν έχουμε ζητήματα να συντονίσουμε, αλλά οι ε, προτεραιότητες μας είναι οι προσεγγίσεις είναι διαφορετικές. Έχουμε την πολιτική μας, έχουμε τα κονδυλιά μας, υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά το τι κάνουμε, ποια είναι η φιλοσοφία μας και τι κάνουμε συγκεκριμένα. Έχουμε προβλήματα όσον αφορά το να λάβουμε τις ανάλογες πληροφορίες από τους Τούρκους συναδέλφους μας. Η προσέγγιση τους στα ζητήματα αυτά είναι διαφορετική. Και παρά το ότι υπάρχει πολύ καλή συνεργασία στο επίπεδο ΥΠΑ της εκπροσώπου και Υπουργών Εξωτερικών, πρέπει να ε, δούμε τη συνεργασία που θα μας επιτρέψει να εργαστούμε στο επίπεδο των προγραμμάτων ε, επιτόπου. Και Γι' αυτό χρειάζονται οι κατάλληλες συνθήκες. Όσον αφορά τις οικονομικές ε, μεταρρυθμίσεις. Η οικονομία ήταν πάντα τμήμα των σχέσεων μας με την νότια γειτονιά μας. Αν δείτε το σχέδιο δράσης πάντα θα βρείτε ένα σημαντικό τμήμα που αφορά τις δημόσιες προμήθειες, φορολογία, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα βασικά δηλαδή οικονομικά κριτήρια που πρέπει να τεθούν σε κάθε χώρα. Σημαίνει αυτό πως πρόσφατα είχαμε την ε, φτάσαμε στα όρια μας το τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε την Αίγυπτο και άλλες χώρες. Όχι, γιατί είχαμε εστιαστεί σε χώρες όπως την Ισία, αλλά και η Αίγυπτος. Η Αίγυπτος αντιμετωπίζει άμεσες οικονομικές ε, προκλήσεις με σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Και πολλά χρήματα πηγαίνουν ειδικά στο να, μείνει, να μείνουν οι νέοι στις ε, περιοχές τους και να μην πάνε στις πρωτεύουσε ή να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. <laughs> Ταυτόχρονα το να έχουμε την εντολή να ξεκινήσουμε μια νέα ε, συμφωνία ελεύθερου η οποία θα μας βοηθήσει ε, όσον αφορά την οικονομική πολιτική της χύψη χώρας. Είμαστε, έχουμε την δυνατότητα να δώσουμε τα δισεκατομμύρια που απαιτεί ο προπολογισμό της ε, Αιγύπτου. Όχι. Γι' αυτό και στενή συνεργασία με τους G8, G20 όπου έχουν γίνει κάποιες υποσχέσεις και στήριξη όχι μόνο από ευρωπαϊκά αλλά και άλλα ε, διεθνή χρηματοδοτικά μέσα. Αλλά ξέρετε, η Κομισιόν δεν έχει τα μέσα να αντιμετωπίσει όλες τις ε, προκλήσεις ε, ειδικά αυτού του μεγέθους. Τώρα, αυτό το οποίο βεβαίω είναι άμεσο και οι αλεπικαλύψεις που υπάρχουν επί τόπου είναι κάτι το οποίο μας ανισχύει, αλλά γι' αυτό υπογράψαμε την συμφωνία με το Συμβούλιο της Ευρώπης για να χρηματοδοτούμε εμείς τα δικά του έργα και να μην υπάρχει αυτή η αλληλεπικάλυψη. Αλλά να στηρίζουμε ένα στον άλλον. Τώρα όσον αφορά τα εθνικά ενδεικτικά προγράμματα έχω δηλώσει επανειλημμένα στην Επιτροπή σας πώς είμαι στη αυσή σας να έρθω όποτε θέλετε να σας εξηγήσω το πώς άλλαξαν τα εθνικά ενδεικτικά προγράμματα, πώς ε, πέρσι την Άνοιξη φροντίσαμε να υπάρχει συμβατότητα μεταξύ εθνικών ενδεικτικών προγραμμάτων και της νέας πολιτικής της γειτονίας. Αυτά είναι ήδη επιτάπτως και επί τη ευκαιρία πολλή δουλειά έχει γίνει, πολλοί πόροι ε, έχουν πάει για να ανταποκριθούν στις προτεραιότητες των χωρών που είναι σε αυτή τη διαδικασία μετασχηματισμού. Είμαι τώρα για μια επίσκεψη από τα κοινοβούλια αυτών των χωρών. Θα το σκεφτούμε οπωσδήποτε. Ε, φοιτητική βίζα. Ναι, ακριβώ αυτό είναι το θέμα της ε, συμφωνίας κινητικότητας. Γιατί για πρώτη φορά έχουμε κράτη-μέλη που συμφωνούν πώς μπορούμε να δούμε ε, τη συμφωνία επανεισδοχής και διευκολύνσεις για τη βίζα ταυτόχρονα. Αυτό δεν συνέβαινε πριν από λίγα χρόνια. Οπωσδήποτε όχι. Πριν από ένα χρόνο δεν υπήρχε κώδικας θεωρήσεων που θα μας επιτρέψει να είμαστε πιο ευέλικτοι όσον αφορά τις ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων όπως φοιτητέ. Η Αλγερία. Δεν ξέρω εάν είπα πως είμαι υπερήφανος για το ότι λάβαμε πρόσκληση να παρατηρήσουμε τις εκλογές. Αλλά αν με ρωτήσατε πώς αντιλαμβάνομαι την πρόοδο στην Αλγερία σε σχέση με την πρώτη μου επίσκεψη, ναι, είμαι υπερήφανος για αυτό το οποίο έχουν γίνει στην Αλγερία. Κάθε χώρα έχει τη δική της πορεία. Πράγματι, οθήθηκαν αρκετοί σημαντικοί νόμοι και αυτή είναι η αρχή της διαδικασίας Σωστά λέτε πως η συνέλευση η οποία τους ψηφίζει είναι η ίδια, αλλά θα γίνουν εκλογές. Και μας ε, κάλεσαν να παρατηρήσουμε αυτές τις εκλογές με ένα στόχο. Δεν θα μας είχαν προσκαλέσει εάν ε, αυτές οι εκλογές... Ε, υπέκρυπταν διάφορα παιχνίδια εμείς θα πάμε εκεί και θα πούμε το εάν αυτές οι εκλογέ είναι πράγματι ελεύθερες και δίκες. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και βεβαίως ε, ε, ναι, με να συναντάω την κοινωνία των πολιτών όπου πάω. Δεν χρειάζεται. Εγώ τη συναντάω παντού ούτω ή άλλω. Και θα συνεχίσω να το κάνω. και θα προετοιμάσω για την επιτροπή σας έναν κατάλογο της οικονομικής βοήθειας και της βοήθειας γενικώ. Ε, και αυτό ίσως ε, θα μπορούσε να μας απασχολεί σε επόμενες ε, συζητήσεις στο ζήτημα, στο ζήτημα αυτό και στο δεικτικό πρόγραμμα γιατί θα γίνει μέχρι το 2013. και για το αν θα εφαρμόσουμε αυτή την αρχή περισσότερα για περισσότερα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους συνάδελφοι, ιδιαίτερα τους εθνικούς βουλευτάς. Σας ευχαριστώ και σας καληνυχτίζω. No, you read it. Seven down, seven down. Seven down, yeah. Seven down. That's beautiful and then Billy, like Willy Brandt. Yes, exactly. the, the Yeah, half an hour ago. Ein Mädchen oder ein... Mädchen, wieder ein Mädchen, hier wie drei Mädchen. Der Name Bruch stirbt aus. Ah, ja. So, Kolleginnen und Kollegen. οι συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Έχουμε μόνο 45 λεπτά για την επόμενη συνεδρίαση, αλλά θα ήθελα να υποδεχτώ τον Υπουργό Εξωτερικών της Δανίας, τον Βίλι Σέρνταλ, να τον ευχαριστήσω για το ότι ήρθε εδώ πέρα να μας ενημερώσει. Νομίζω πως πρέπει να είμαστε σύντομοι, περιεκτικοί να ασχοληθούμε με κάποια ουσιαστικά ζητήματα. ήθελα... μπορούσε να είναι και το Ιράν. Αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Υπουργό να κάνει μια σύντομη εισαγωγή και λόγω του χρόνου ο οποίος πιέζει ο κάθε μιλητής θα μιλήσει για ένα λεπτό για να μπορέσουν να μιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Συμφωνείτε? Ωραία. Κύριε Υπουργέ, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια για τα νέα σας καθήκοντα ε, Πρόεδρο της Επιτροπής. Θα ήθελα να ξεκινήσω τονίζοντας πως δεν έχω έρθει εδώ πέρα με την εθνική μου ιδιότητα, εκπροσωπώ την είπατε εκπρόσωπο για να σας ενημερώσω για κάποια πράγματα. Ο κύριος Βάμεν, ο Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, θα σας, παρουσιάσει αμέσως μετά μια οπτική της ε, Δανίας. Χτες είχαμε λοιπόν ένα πολύ ενδιαφέρον Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, συζητήσαμε σημαντικά ζητήματα και λάβαμε αποφάσεις κλειδιά. Για πρώτη φορά συμμετείχε και η Κροατία στο Συμβούλιο ως παρατηρητής μία μέρα μόλις μετά το επιτυχές δημοψήφισμα. Το πιο κατεπήγον ζήτημα ήταν το Ιράν, το οποίο ήταν άρα και πρώτο στην ημερήσια διάταξη. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου τα συμφωνήσαμε, καθώς και ένα σημαντικό νέο πακέτο κυρώσεων, το οποίο στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στο Ιράν, συμπεριλαμβάνονται εκεί πέρα σημαντικές απαγορεύσεις για την εισαγωγή πετρελαίου από το Ιράν και η Κεντρική Τράπεζα του Ιράν και η Τράπεζα Τεχράτ ε, εξακολουθούν να αποτελούν ακόμα αποδεκτούς εμπορικούς εταίρους. Επίσης υπάρχουν ρήτρες αναθεώρησης οι οποίες θα επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να επανεξετάσει την κατάσταση σε λίγους μήνες για να διασφαλιστεί η ε, ασφάλεια ενεργειακής παροχής ε, των κρατών μελών. Ελπίζουμε επίσης αυτό να έχει ένα αντίκτυπο έτσι ώστε και άλλες χώρες να μπορέσουν να μας ακολουθήσουν. Οι κυρώσεις αυτές βεβαίως δεν είναι αυτός σκοπός. Ο στόχος μας παραμένει μια διπλωματική λύση. Θα ήθελα να τονίσω εδώ την ξεκάθαρη δέσμευση της Ένωσης για την διπλή αυτή προσέγγιση. Οι διπλωματικές μας προσπάθειες συνεχίζονται και εξακολουθούμε να αναμένουμε μια σαφή επίδραση από το Ιράν στις προτάσεις μας. Το Ιράν τώρα πρέπει να κάνει μια επιλογή, επιθυμεί το διάλογο πρέπει να δείξει πως είναι έτοιμο να ε, κάνει μαζί μας επικοδομητικές συνομιλίες χωρίς ε, ε, προαπαιτούμενα. Κατόπιν ασχοληθήκαμε με τη Βερμανία Μιανμάρ και καλωσορίσαμε τις εξαιρετικές πολιτικές εξελίξεις εκεί. Συμφωνήσαμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιδράσει θετικά και γρήγορα ως ένα πρώτο βήμα θα αρθεί η απαγόρευση θεωρήσεων για τα μέλη της κυβέρνησης. Επίσης προετοιμαζόμαστε να υποστηρίξουμε την ε, μετάβαση και το λαό της Βυρμανίας Μιανμάρ. Ο Επίτροπος Πίμπαλξ ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα 150 εκατομμυρίων υποθέτω ευρώ μέχρι το 2013 και βεβαίως αναμένουμε το τι μπορεί να γίνει για να είναι επιλέξιμη η Βερμανία, Μιανμάρ για την πρωτοβουλία για εμπόριο σε όλους τους τομείς πλην των όπλων. Η δε ε, κυρία Άστον είχε συναντηθεί ούτως ή και με την αν Σαν τον Απρίλιο μετά τις εκλογές. Το Συμβούλιο λοιπόν καλωσορίζει τις αλλαγές που έλαβαν χώρα και αυτή είναι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα όσον αφορά την κρίση στην Συρία που ήταν το επόμενο θέμα μας. Συμφωνήσαμε πως η κατάσταση ήταν άσχημη και χειροτερεύει. Ο Αραβικός Σύνδεσμος αποφάσισε την Κυριακή να ενισχύσει την αποστολή παρατηρητών. Η ύπατη εκπρόσωπος μας ενημέρωσε για το ότι μίλησε με το Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου και προσέφερε την πλήρη στήριξή μας στις προσπάθειές του μέσω ε, της σύστασης μιας ομάδας παρόμοιας με την ομάδα του Καΐρου στη, για τη Λιβύη, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Αραβικός Σύνδεσμος και ε, άλλες χώρες του ΟΑΣΕ θα συμμετέχουν. Καλώς ορίσαμε λοιπόν την πρωτοβουλία του Αραβικού Συνδέσμου της 23ης ε, Φεβρουαρίου και την στήριξη στην πολιτική λύση. Ζητάμε και πάλι τερματισμό της βίας, παρατηρητές του Αραβικού Συνδέσμου να μπορέσουν να εργαστούν ελεύθερα να μπορέσουν να στηρίξουν το λαό και οτιδήποτε μπορεί να γίνει για να επιτύχουμε μια ειρηνική μετάβαση. Επιπλέον αυξήσαμε την πίεση στο καθεστώς με επιπλέον κυρώσεις ε, κατά νέων ατόμων και επιχειρήσεων ένα μεγάλο αριθμό ατόμων και επιχειρήσεων. το ζήτημα κατόπιν της Σερβίας και του κατά πόσο θα είναι υποψήφια χώρα θα τεθεί στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της 28 Φεβρουαρίου. Εν ώψη αυτή της συζήτηση έγινε μια πάρα πολύ καλή συζήτηση για την τρέχουσα κατάσταση καθώς επίσης και τις σχέσεις Σερβίας-Κοσφοπεδίου. Όταν λήφθη η απόφαση του Δεκεμβρίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είχαν τραυματιστεί στρατιώτες της ΚΕΙΦΟΡ από κράτη-μέλη, κάτι το οποίο δεν μπορούσαμε να γνωρίσουμε. Έχει επιτευχθεί τώρα λογική πρόοδος έκτοτε, αλλά η περαιτέρω πρόοδος εξαρτάται από την προθυμία και των δύο πλευρών να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Εμείς συμφωνήσαμε πως ελπίζουμε να δούμε και τη Σερβία και το Κωσυφοπαίδιο να προχωρήσουν στις σχέσεις τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά όσον αφορά την περιφερειακή συνεργασία. Στο μεσημεριανό γεύμα συζητήσαμε την Αίγυπτο και την ειρηνευτική διαδικασία. Όσον αφορά την ειρηνευτική διαδικασία, ανταλλάξαμε απόψεις για το πώς θα συνεχιστούν οι απευθείας διαπραγματεύσεις. Η ύπατη εκπρόσωπος αναφέρθηκε στις ε, συμφωνίες ε, με την Ιορτανία και σήμερα θα επισκεφθεί το Ισραήλ και σκοπεύει να συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου, τον Υπουργό Εξωτερικών Λίμπερμαν, ε, τον Πρόεδρο Αμπάς και τον Πρωθυπουργό των Παλαιστινίων. Και υιοθετήσαμε συμπεράσματα του Συμβουλίου που επιβεβαιώνουν την πάγια θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους επικισμούς. Τέλος, υιοθετήσαμε μια θέση για έναν νέο ειδικό αυσταλμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ανδρέας Ράινιγκερ, όσον αφορά την Αίγυπτο. Χτες ε, η Λαϊκή Συνέλευση, το Κοινοβούλιο δηλαδή, συνεδρίασε για πρώτη φορά, είπατε εκπρόσωπος, ε, ξέρω σε μια ανακοίνωση λέγοντας πως ελπίζουμε το Κοινοβούλιο να οδηγήσει σε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του λαού για οικονομικά, και κοινωνικά δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες. Αναμένουμε λοιπόν το Μεγάλο Συμβούλιο της ΣΟΥΡΑ, τη λεγόμενη η οποία θα ξεκινήσει 29 Ιανουαρίου. Αποδίδουμε μεγάλη σημασία στη μετάβαση στην πολιτική εξουσία των στομότερων δυνατών για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του Αιγυπτιακού λαού έχει μεγάλη σημασία οι αρχές να τηρήσουν την δέσμευσή τους να γίνουν προεδρικές εκλογές μέχρι το τέλος του Ιουνίου φέτος. Μετά το φαγητό συζητήσαμε την ανησυχητική κατάσταση στη Λευκορωσία και τα επόμενα βήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρχε ευρεία συνένεση στο ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν λόγια αισιοδοξία, οπότε συμφωνήσαμε στο να επεκτείνουμε τα κριτήρια κυρώσεων, ε, στο να συμπεριλάβουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και ανθρώπους που είναι κοντά στο καθεστώς. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε επ' αυτών για να συμπεριλάβουμε περισσότερα ονόματα στην απαγόρευση βίζας. Επίσης συζητήσαμε το πώς θα μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή με τους ανθρώπους της Λευκορωσίας μέσω Τη κοινωνία των πολιτών πρέπει να τεθούν τα θεμέλια για τη μελλοντική δημοκρατική Λευκορωσία και θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό το Φεβρουάριο. Οι Υπουργοί ανησυχούσαν για τις σχέσεις μεταξύ Σουδάν και Νοτίου Σουδάν. Εκούσαμε μια έκθεση από την κυρία Γεωργίευα, την Επίτροπο, την Επίτροπο η οποία ανέφερε τα κυριότερα ζητήματα και βεβαίω οι υπουργοί συζήτησαν ακόμα τα εκκρεμή ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών. Στόχο είναι δύο χώρε που θα συμβιώνουν ειρηνικά. Ανησυχούμε ιδιαίτερα για τι συγκρούσει στον Γαλαζιονίλο, στο Σουδάν που έχουν καταλήξει σε μεγάλο αριθμό εκτοπισμένων. Ζητάμε λοιπόν από την κυβέρνηση του Σουδάν να επιτρέψει η ανθρωπιστική πρόσβαση σε όσου την έχουν ανάγκη. Επίση, ανησυχούμε για τι βίαιε συγκρούσει μεταξύ κοινοτήτων στο νότιο Σουδάν. Καλωσορίζουμε το επιτυχημένο έργο της ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράση την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη σε μια κοινή στρατηγική για τον Νότιο Σουδάν με κινητοποίηση πάνω από 800 εκατομμυρίων ευρώ υιοθετήθηκαν συμπεράσματα του Συμβουλίου. Στα διάφορα συζητήθηκαν τα συγκλονιστικά γεγονότα στην Νιγηρία και σε μελλοντικέ επαφέ με την κυβέρνηση της Νιγηρίας θα συζητήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε από αυτό. Όσον αφορά το ευρύτερο ζήτημα της ε, Άνοιξη σκίας και της ελευθερία άσκηση της θρησκεία, είπαμε πω είναι κακό πράγμα η διώξη των θρησκευτικών μειονοτήτων. Αυτά ήταν τα θέματα που συζητήσαμε χθε στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Εννέα ομιλητέ και ομιλήτριε. Νομίζω πρέπει να κλείσουμε τον κατάλογο. Γιατί μετά θα έχουμε κι άλλον υπουργό. Πρώτα οι συντονιστές ένα λεπτό ο καθένας. Σαλαφράγκας. Ευχαριστώ Πρόεδρε και Υπουργέ, σας καλωσορίζω, καλή επιτυχία στο εξάμεινο της Προεδρίας σας και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ε, ενημέρωση που μας κάνατε σχετικά με το χθεσινό συμβούλιο. Αλλά σε λίγο θα έρθει και ο συνάδελφό σα. Τώρα, σε ό,τι φορά τι κυρώσει κατά του Ιράν, αυτέ οι κυρώσει και το εμπάρκο πετρελαίου θα είναι αποτελεσματικέ και αν δεν είναι αποτελεσματικέ, τι περιθώρια υπάρχουν για επιμέρου κυρώσει. Τώρα, εκεί στην Ανατολή, να συγχαρώ για τον διορισμό του προσώπου μα. Πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το αίτημα της Παλαιστίνης για να γίνει μέλος ε, του ΟΗΕ έχει εναρμονισμένη θέση και τέλος Συρία. Στο τελευταίο σημείο των συμπερισμάτων του Συμβουλίου καλείται τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να αναλάβουν τις ευθύνες τους σε αυτό το όργανο του ΟΗΕ. Θεωρείται ότι είναι εφικτό. Υπενθυμίζω ότι είμαστε 10 χρόνια από την ε, επέμβαση του Ιράκ στο Ιράκ συγγνώμη, και το Συμβούλιο Ασφαλείας θα μπορούσε να λάβει επιτέλου μια απόφαση σοβαρή για το τέκτανο της Συρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την παρουσία σας. Έχω δύο ερωτήσεις. Πρώτον για τη Σερβία. Πώς θα λέγατε ότι είναι το κλίμα εκεί. Οι αποφάσεις που αναμένουμε το Μάρτιο γίνονται κατανοητές ως σημαντικές για την περιφέρεια και το μέλλον της χώρας. Νομίζετε ότι βελτιώνονται τα πράγματα σε σύγκριση με το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Δεύτερο για την Πελαρούς. Πέρα από την παράταση των κυρώσεων, πώς βλέπετε τη συζήτηση των εκπροσώπων των χωρών μελών για την Πελαρούς. Αναγνωρίζουν ότι δεν υπάρχουν αποτελέσματα μέχρι τώρα ή υπάρχει καμία καινούργια ιδέα πώς να προσεγγίσουμε την κοινωνία της Μπελαρούς για να έχουμε οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Μήπως η κατάσταση έχει χειροτερέψει αντί να βελτιωθεί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γέλος και θυμίδια. Καλωσορίζω τον Υπουργό στην Επιτροπή μας εξ ονόματος της ομάδας μου και πόσο μάλλον που είναι και μέλος της πολιτικής μας οικογένειας. Στη χθεσινή συνεδρία των Υπουργών Εξωτερικών για τα Βαλκάνια και το Κωσυφοπαίδιο είπατε ότι χρειάζεται καλή θέληση και από τις δύο πλευρές και το πρωί με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε η έκθεσή μου για το Κωσυφοπαίδιο που όπου έλεγα ότι πρέπει τα κράτη-μέλη να το αναγνωρίσουν και να ζητήσουν από τη Σερβία να προχωρήσει σε αυτή τη συνεργασία αν θέλει να ε, προχωρήσει στην οδό της εντάξεως ή μάλλον της υποψηφιότητας. Εσείς πώς το βλέπετε. Ξέρω ότι ο διάλογος μεταξύ Σερβίας και Κωσυφοπεδίου γίνεται προσπάθεια να ενισχυθεί, αλλά οι υπουργοί τι λένε. Η Δανική Προεδρία είναι σαφής ότι είναι υπέρ της διεύρυνσης. Θέλετε να ανοίξουν περισσότερα κεφάλαια με την Τουρκία Ευχαριστώ Πρόεδρε κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να διαφωνήσω για την απόφαση που λήφθη αναφορικά με το εμπάργκο προς το Ιράν. Είναι μια απόφαση ανεύθυνη και δεν νομίζω, ότι η επόμενη άλλη λύση θα ήταν η πυρηνικοποίηση, αν θέλετε, στην, της περιοχής. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαδραματίσει ένα διαφορετικό ρόλο να προωθήσει μια διεθνή συνθήκη που θα απαγορεύει και θα καταστρέφει όλο το, τον πυρηνικό εξοπλισμό. Αυτό, διαφορετικά είμαστε υποκριτές διότι άτομα, ε, συγγνώμη, κράτη τα οποία έχουν δυνατότητα να καταστρέψουν 7 φορές τον πλανήτη με τα όπλα τους να απαγορεύουν σε άλλα κράτη να κατέχουν την πυρηνική ενέργεια. Εγώ είμαι κατά της ε, πυρηνικής ενέργειας, κατά των εργοστασίων ε, παραγωγής ηλεκτρική ε, ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνικά. Πάντως νομίζω ότι το μέτρο αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για μια περιοχή όπως αυτή της Μέσης Ανατολής θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραγωδία εάν δεν ενεχθεί. Ξέρετε ότι τα προβλήματα τα πληρώνουν οι λαοί και όχι οι κυβερνήσεις. Θεωρώ η απόφαση είναι εσφαλμένη και καταλήγω Πρόεδρε να ζητήσω την αναγνώριση της, του Παλαιστινιακού κράτους. Thank you, President. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ. Χθες ε, διαβάσαμε κάποιες ειδήσει εδώ, εδώ, εδώ μπροστά σας Το Ιράν εξεπλάγει που η Ευρωπαϊκή Ένωση κράτησε μια ομόφωνη θέση. Θα πρέπει κάτι τέτοιο να το βλέπουμε πιο συχνά και ελπίζουμε να έχει σημαντικές συνέπειες. Ε, θα ήθελα να γνωρίζω ότι πραγματικά πιστεύετε Ειδικά με τα, ε, με τα κίνητρα προκειμένου το Ιράν να μπορέσει να βγει από την κατάσταση που βρίσκεται τώρα, που βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο κατά κάποιο τρόπο. Θεωρούμε ότι η κατάσταση αυτή είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, όπου οι ηγέτε όπω η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενεργήσουν με την απόλυτη υπευθυνότητα. Θα πρέπει να ε, δρούμε ανεξάρτητα από τις ΗΠΑ, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το Ιράν. Παράλληλα να αναφερθώ στα παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνεχίζουν να γίνονται στο Ιράν. Σε ό,τι αφορά το γεωπολιτικό ζήτημα, ε, ακούσαμε ότι, θα, ότι υπάρχουν περαιτέρω, προσπάθει, περαιτέρω συλλήψεις ε, δημοσιογράφων κλπ συμφωνήσουμε τόσο είπε να συνάδελφος Σαραφράν για τη Συρία. Δεν μπορούμε να καθόμαστε με ψευρωμένα τα χέρια. Θα πρέπει να βρούμε κάποιες ε, επιλογές ε, όπως ε, να καλέσουμε τις οικονομικές ελίτ ή να ζητήσουμε από τις αγορές να λάβουν ξεκάθαρες αποφάσεις. Ευχαριστώ. Λυπάμαι. Χαίρομαι, Πρόεδρε, που συζητιέται επιτέλους η Μέση Ανατολή, αν και δεν καταλαβαίνω γιατί ακόμα συζητάμε τις ανοησίες του κουαρτέτου. Ο νέος ειδικό απεσταλμένος υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργήσει ακόμα περισσότερη σύγχυση από ό,τι πριν. Και δεν χρειάζεται ένας ακόμη επιτόπου. Έπειτα θα ήθελα κάποιες περισσότερες πληροφορίες για την αντίδραση του Συμβουλίου λόγω της αλλαγής πολιτικής της Αιγύπτου και των προβλημάτων στη Συρία. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρον ο κόσμος σε αυτήν τη φάση που ζούμε και σε τόσο πολλά μέρη του κόσμου. Πρώτον για την Παλαιστίνη και την ένταξή της ή την υποψηφιότητά της στον ΟΗΕ Αν με ρωτάτε αν οι Υπουργοί Εξωτερικών ήταν αισιόδοξοι και πίστευαν ότι θα κατέληγε αυτό σε κανένα αυτό αποτέλεσμα, θα σας έλεγα όχι. Είτε λοιπόν οι Παλαιστίνοι θέλουν να λυθεί το θέμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ Ξέρουμε τι θα γίνει αν τεθεί αυτό εκεί. Τίποτε. Και η άλλη δυνατότητα είναι να το θέσουν στη Γενική Συνέλευση. Τότε θα ψηφιστεί η ενίσχυση του καθεστώτος των Παλαιστινίων, αλλά δεν ξέρω αν θα το κάνουν. Αν θέλουν να το κάνουν, τότε οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες θα υποστηρίξουν την πρόταση αυτή νέου καθεστώτος για την Παλαιστίνη στον ΟΗΕ. για την απόφαση της Σερβίας. Όλοι νόμιζαν ότι τα πράγματα είχαν αλλάξει από την προηγούμενη φορά που συζητήθηκε το θέμα τον Δεκέμβριο και ότι κινήθηκαν προς τη σωστή κατεύθυνση. Ακόμη όμως πρέπει να γίνουν κι άλλα. Και για το κοσυφοπέδιο πρέπει βέβαια να βελτιωθούν οι σχέσεις με τη Σερβία. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματα και ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να λυθούν. Αλλά προσπαθούμε να κάνουμε γενναία και θαραλέα βήματα για πρόσβαση στην Ένωση. Και λέω προσωπικά και ότι ελπίζω τον Μάρτιο, Φεβρουάριο-Μάρτιο, να είμαστε σε θέση να φέρουμε τη Σερβία κοντύτερα στην Ένωση. Το κλίμα είναι καλό λοιπόν μεταξύ νομίζω όλων των χωρών. Το θέμα είναι όμως πόσες δηλώσεις θα... Α, ε, τι προϋποθέσεις πρέπει να υπάρξουν που να τις πραγματοποιήσει η Σερβία αλλά και οι υπόλοιποι. Για το Ιράν Όσοι επικρίνουν και λένε ότι δεν θα έπρεπε να είχαμε κάνει αυτό το πράγμα, θα έλεγα ότι τρία πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Πρώτον, τίποτα. Σε αυτή την περίπτωση όμως υπάρχει ο κίνδυνος αν πιστέψουμε την έκθεση της Επιτροπής Πυρηνικής Ενεργείας ότι το Ιράν σε 1,5 χρόνο θα είναι πυρηνική δύναμη, αν γίνει κάτι τέτοιο τότε θα διαδοθούν στη Μέση Ανατολή τα πυρηνικά όπλα γιατί και άλλες χώρες θα θέλουν. Αυτό είναι απειλή για όλους μας. Η άλλη δυνατότητα είναι να χρησιμοποιήσουμε στρατιωτική γλώσσα. Δεν είναι καλό πράγμα αυτό. Και τρίτη και μόνη η δυνατότητα είναι να συνδυάσουμε τις κυρώσεις με τη δυνατότητα πολιτικών διαπραγματεύσεων. Αυτό ακριβώς θέλουν να κάνουν οι Υπουργοί Εξωτερικών. Τέλος για την Αίγυπτο και τη Συρία. Για την Αίγυπτο φαίνεται ότι θα υπάρξει κυβέρνηση. Δεν ξέρουμε πότε ή τι ποιο ρόλο ακριβώς θα παίξει η μουσουλμανική αδελφό της. Αλλά νομίζω ότι θα ήταν λάθος να κρίνουμε τα πολιτικά αυτά κόμματα επιφανειακά. Πρέπει να τους κρίνουμε από τις πράξεις τους, όχι από τα ονόματά τους. Η Αίγυπτος νομίζω θα εφαρμόσει τις συμφωνίες που έχουμε ήδη συνάψει εκεί Ίσως να μην υπάρξει καμιά τεράστια αλλαγή, αλλά δεν είμαι και βέβαιος, στην εξωτερική πολιτική της Αιγύπτου. Το σημαντικότερο είναι νομίζω ότι είμαστε παρόντες εκεί και άρα οι προσπάθειες των θαραλέων νεαρών που είδα και ο ίδιος στην πλατεία Ταχρήρ γιατί είδα και ένα νέο περίπου 30 ετών που μου είπε και εγώ βοήθησα και ήταν περήφανη η μητέρα μου αν και ο πατέρας μου είναι στρατηγός. Αυτό νομίζω δείχνει πόσες ελπίδες είχαν γεννηθεί πέρυσι πρέπει να συνεχιστεί αυτό, να παραμείνουμε παρόντες εκεί για να μπορέσουν να διατηρήσουν αυτήν την ελπίδα ότι θα υπάρξει η δημοκρατική μετάβαση. Δεν είναι ποτέ ευθεία αυτή η οδός. Θα υπάρξουν και οι και πράγματα που δεν θα μας αρέσουν, αλλά η καλύτερη εγγύηση που μπορούμε να δώσουμε ή τουλάχιστον βοήθεια είναι να παραμείνουμε εκεί παρόντες στην Αίγυπτο μάλιστα. Για τη Συρία νομίζω ότι η σημαντική βοήθεια που μπορούμε να δώσουμε θα ήταν να οδηγήσουμε τα πράγματα στην οδό της μη βίας, της αποφυγής της βίας να καταδικαστούν οι βιαιοπραγίες που αυτή τη στιγμή είναι τεράστιες, πάνω από 5.000 σκοτώνονται. Πολλοί χάνονται και πολλοί φυλακίζονται. Αυτό είναι πολύ σκληρό, τόσο σκληρό που πρέπει σαφώς να καταδικάσουμε αυτά που γίνονται σήμερα στη Συρία. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα η κυρία Κρόνμπεκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να σχολιάσω λίγο τη διπλή οδό που αναφέρατε, δηλαδή κυρώσεις και διαπραγματεύσεις. Πρέπει όμως να εξισορροπηθεί το ένα με το άλλο. Ο κίνδυνος των νέων κυρώσεων είναι ότι δεν συνοδεύονται από νέες προτάσεις για διαπραγματεύσεις. Η Κατερίνη Άστον περιμένει από τους Ιρανούς να διαπραγματευτούν χωρίς προϋποθέσεις. Και η ίδια έθεσε προϋποθέσεις. Το Ιράν δηλαδή να ακολουθήσει τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Πού βρίσκεται εδώ η διαπραγμάτευση και πώς αναμένει το Συμβούλιο από την Ιρανική κυβέρνηση αφού την έχει βάλει στη γωνία, εκείνοι να μην θέτουν όρους και εμείς να θέτουμε, να ανταποκριθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την παρουσίαση. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας και να σας ε, ρωτήσω σχετικά με το ζήτημα των δικαιωμάτων ε, που σε παρουσίασε η Βαρονή Άστον στο κρατημένο δέξη στο Κοινοβούλιο για βελτίωση των μέσων που έχουμε διάθεσή μας. κράτη-μέλη δουλεύουν πάνω σε αυτά τα ζητήματα και εμείς στο Κοινοβούλιο. Θα θέλω να ακούσω από εσά από την Προεδρία Πιστεύετε ότι θα ήταν δυνατόν στο τέλος της Δανικής Προεδρίας να έχουμε ε, έχουμε μια ενίσχυση των ε, συμφωνίων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να τονίζουμε ότι για μας το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερη σημασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και σας και τον Υπουργό. Εγώ είμαι πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου για σχέσεις με το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο. Και θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για το Παλαιστινιακό. Είπατε ότι οι διαπραγματεύσεις, οι συζητήσεις έγιναν σε ένα γεύμα. Προβλέπεται όμως κάποια πρόοδος για τις σχέσεις Παλαιστινίων και Ισραηλινών με βάση τις συζητήσεις που γίνονται. Καταφέρατε να υπάρξει συμφωνία σε ολόκληρη την Ένωση για κυρώσεις και διαπραγματεύσεις με το Ιράν αλλά φαίνεται ότι δεν έγινε καμία προσπάθεια να ακολουθηθεί η ίδια μέθοδος και στη Μέση Ανατολή. Πράγματι υπάρχουν κατάφορες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ μέρους του Ισραήλ, ακόμη και κατά παιδιών. Εκατοντάδες φυλακίζονται, βασανίζονται, κρατιούνται στην απομόνωση ανακρίνονται από στρατιωτικούς παιδιά, τη απουσία των γονέων τους κλπ. Πρέπει λοιπόν να επανεξισορροπηθεί η στάση της Ένωσης. Το αναλαμβάνετε εσείς αυτό σαν καθήκον της Προεδρίας. Ευχαριστώ. Η κυρία Γόμης που είναι και η συγγήτρια για τη Λιβύη. Ναι αλλά δεν θα θέσω ερώτημα για τη Λιβύη αλλά για το Ιράν. Είμαι υπέρ των κυρώσεων και υπέρ των διαπραγματεύσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Λοιπόν, στις κυρώσεις που έχουν αποφασιστεί, σκεφτήκατε να δώσετε ένα σαφές μήνυμα προς τις τράπεζες της Ένωσης που στο παρελθόν τουλάχιστον κατάφερναν να παραβιάσουν τις κυρώσεις αυτές. συζητήσατε καθόλου για την Ουκρανία την πιθανότητα απελευθέρωσης της κυρίας Τιμόσενκο. Και σε μια χώρα που είναι η, πολυπληθε, η δεύτερη πολυπληθέστερη της Αφρικής, την Αιθιοπία δηλαδή, δύο Σουηδοί δημοσιογράφοι συνελήφθησαν, πέντε Ευρωπαίοι συνελήφθησαν, έγιναν τεράστιες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χειραγώγηση των εκλογών θα συνεχίσετε να μην τα βλέπετε όλα αυτά. Ο κύριος Σούλτς τελευταίος. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Μια ερώτηση για τη Λευκορωσία. Είπατε πως θα το ξανασυζητήσετε το θέμα το Φεβρουάριο και τα κριτήρια α, των κυρώσεων θα διευρυνθούν. Γνωρίζουμε όμως πως Μέχρι τώρα το μπλοκάρισμα λογαριασμών και ταξιδιού δεν είχε αποτέλεσμα. Οπότε η επέκταση αυτών των ε, κυρώσεων δεν ε, είναι παρά μόνο το καθεστώς Λουκασέγκο να επιβάλλει σκληρότερη καταπίεση. Θα επιβάλλεται στοχευμένες κυρώσεις. Κοιτάξτε, εγώ τώρα δεν είμαι υπέρ τόσο των οικονομικών κυρώσεων, αλλά αν ξέρει κανείς την οικονομική δομή όπου οι περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις είναι στα χέρια του κράτους, δηλαδή της κλίκας του Λουκασέγκο και πάνε τα κέρδη κατευθείαν στις τσέπες τους, τότε νομίζω μπορεί να βοηθήσουν οι οικονομικές ε, κυρώσεις. Ε, νομίζω πως μόνο δύο-τρεις χώρες εμποδίζουν ε, το Συμβούλιο. Υπάρχει η δυνατότητα, ξέρω εγώ, να δώσουμε και κάποια αποζημίωση, όπως στην περίπτωση της Λετωνίας. Σας ευχαριστώ και πάλι. Θα ξεκινήσω από την αρχή, ε, δηλαδή από το Ιράν. Το ερώτημα ήταν πώς μπορείτε να λέτε πως είναι πιθανό πως θα λειτουργήσουν αυτές οι κυρώσεις στο Ιράν για ποιο λόγο δηλαδή, νομίζω για δύο-τρεις λόγους. Το ένα είναι πως το καθεστώς του Ιράν δεν συμφωνεί για το ποιο τίμημα είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν. Ο ένας λόγος είναι αυτός. Ο άλλος είναι πως οπωσδήποτε δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιες κυρώσεις και να πλήττονται μόνο όσοι είναι κοντά στο καθώς. Το δεύτερον είναι πως θα πλήξουν και τον ε, πληθυσμό και μέρος Ευρώπης. Είναι αδύνατον να επιβάλλουμε κυρώσεις που δεν ε, ε, χτυπάνε καθόλου εάν είναι πραγματικά να λειτουργήσουν. Οπότε ήδη η Ιρανική οικονομία συρρυκνώνεται. Οι κυρώσεις που επιβάλλουμε είναι τόσο ουσιαστικές ώστε θεωρούμε πως ε, θα ε, εξαναγκάσει το, εξαναγκάσουν το Ιράν να επανεξετάσει τα πράγματα. Επίσης, εάν δείτε τις κυρώσεις αυτές ε, και αν ρωτήσει κανείς, μα λειτουργούν ποτέ οι κυρώσεις. Ναι, καμιά φορά λειτουργούν. Χτες ήρθαν κάποιες κυρώσεις επί της Βυρμανίας. Αυτό το κάναμε γιατί λειτουργήσαν. Μπορεί να συζητήσει κανείς βεβαίως πάντα το τι άλλαξε την κατάσταση στη Γερμανία, αλλά εγώ θεωρώ πως οπωσδήποτε και οι κυρώσεις έπαιξαν ένα ρόλο. Το ίδιο και με το καθεστώς της Νοτιοαφρικής Αφρικής επί Απαρτχάιτ. Αλλά όταν επιβάλλει κανεί κυρώσει, σημαντικό είναι το ότι υπάρχουν πολλές χώρες που είναι διατεθειμένες να το κάνουν μαζί, από κοινού. Όχι να φροντίσουμε πως το πετρέλαιο το οποίο ερχόταν στην Ευρώπη το πουλάει το Ιράν αλλού. Τότε δεν κάνουμε τίποτα. Και επίσης να υπάρχει μια εσωτερική αντιπολίτευση στη χώρα με την οποία να μπορούμε να συζητήσουμε. Όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, κάποιες παρατηρήσεις. Πριν από έξι μήνες υπήρξε ένα κοινό έγγραφο με τη Γερμανία για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το συζητήσαμε το Δεκέμβριο, η Υπουργεία Εξωτερικών και κατόπιν τον Μάρτιο στο Συμβούλιο του ΚΙΜΝΕΚ έχουμε δύο ημερήσιες διατάξεις. Η μία αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα συντάξουμε ένα έγγραφο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για τη νέα κυβέρνηση της Δανίας τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πολύ σημαντικά. Ορίσαμε μόλις έναν πρέσβη ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να ληφθεί υπόψη αυτό το ζήτημα. Όσον αφορά δε αυτό το οποίο ρώτησε ο κύριος Ντερόσα ε, για την αισιοδοξία για τη Μέση Ανατολή, είναι δύσκολο να είναι κανείς αισιόδοξο για την εξεύρεση λύσης και είναι κρίμα. Γιατί βεβαίως ε, όλοι οι κάτοικοι της περιοχής χάνουν σε σχέση με τι εξελίξει τη τωρινή βεβαίω. Η Παλαιστίνη είναι προφανές αν δει κανεί την κατάσταση στη Γάζα και τη δική Όχθη, είναι αυτοί που χάνουν περισσότερα, αλλά και το Ισραήλ. Και μια προσωπική παρατήρηση, ε, θεωρώ πως είναι σημαντικό να βοηθήσουμε από έξω ε, να φτάσει η κατάσταση σε ένα σημείο κινητικότητας μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα. Υπάρχει η πιθανότητα, ειδικά η Ευρώπη, να φροντίσει την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη και νομίζω πως είναι σημαντικό να σκεφτούμε το πώς θα φροντίσουμε η Παλαιστινιακή ηγεσία να μην εξασθενήσει την πολιτική διαδικασία. γιατί δεν υπάρχει μια καλύτερη εναλλακτική. Αυτή ήταν όμως μια προσωπική παρατήρηση. Ο κύριος Γκόμες, η κυρία Γκόμες, με συγχωρείτε, με ρώτησε για την κατάσταση της κυρίας Τιμοσένκο. Το συζητήσαμε οι υπουργοί γιατί ξέρετε πως έχουμε τη συμφωνία σύνδεσης. Είναι σημαντικό να τελειώσει η τεχνική πτυχή δεν θα την υπογράψουμε, αλλά πρέπει να τελειώσουμε τις διαπραγματεύσεις και θα πούμε όταν σταματήσετε να ανακατεύετε την πολιτική ε, με τις νομικές διαδικασίες ε, τότε θέλουμε να έχουμε μια καλύτερη σχέση μαζί σας. Αλλά είναι ε, αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ουκρανία μας προβληματίζει και πολύ περισσότερο από αυτό που συμβαίνουν στη Λευκορωσία. Είναι δύσκολο να βρει κανείς μια απλή απάντηση σε αυτά. Η κατάσταση πάει στη λάθος κατεύθυνση. Από την άλλη, δεν θέλουμε να σπρώξουμε την Ουκρανία και τη Λευκορωσία στην αγκαλιά της Ρωσίας. Αυτό είναι το δίλημα που αντιμετωπίζουμε. και προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε όσο δυνατόν καλύτερα. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ήταν μια σωστή παρουσίαση μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην Προεδρία σας και ελπίζουμε να αποδώσει προς όφελος όλων μας.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 Äh, Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να αποδεχτούμε τον Νικολάη Βάμεν, Δανό Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Προεδρεύοντα του Συμβουλίου για το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Θα αναφέρει τις προτεραιότητε της Προεδρίας της Δανίας ειδικά στον τομέα τη πολιτική αλλά και των οικονομικών μέσων. Αναμένουμε λοιπόν την παρουσίασή σας. Έχετε το λόγο. Thank And, uh, first Ευχαριστώ Πρόεδρε, να σας συγχαρώ για την πρόσφατη εκλογή σας. Διακεκριμένα μέλη της Επιτροπής. Με ιδιαίτερη χαρά σας κάνω αυτή την ενημέρωση σήμερα και να κάνω κάποιες αγωγικές παρατηρήσεις αναφορικά με τις προτεραιότητες της Δανικής Προεδρίας. Μετά θα περάσω στην ε, διεύνηση και ε, πολιτική γειτονία και θα θίξω επίσης και το ζήτημα των δικαιωμάτων και ευχαρίστω μετά να ακούσω τις ερωτήσεις σας. Ως εισαγωγή θα ήθελα εντάχει να αναφερθώ στις τέσσερις προτεραιότητες της ε, Δανικής Προεδρίας. Πρώτον, υπεύθυνη Ευρώπη. Δεύτερον, μια δυναμική Ευρώπη. Τρίτον, μια πράσινη Ευρώπη και τέλος μια ασφαλή Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά την πρώτη προτεραιότητα, ε, υπεύθυνη Ευρώπη, είναι ξεκάθαρο ότι θέλουμε να ε, μην υπάρχουν ε, ανισορροπίες στην ευρωπαϊκή οικονομία και αστάθειες. Θα πρέπει να ανταποκριθούμε άμεσα στις ανάγκες που αντιμετωπίζουν κάποιες ε, υπερχρεωμένες ευρωπαϊκές οικονομίες. Χρειάζεται λοιπόν πολιτική βούληση για τήρηση των νέων κανόνων στην ε, οικονομική διακυβέρνηση. Αυτοί είναι κανόνες ε, που θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της Δανικής Προεδρίας. Το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020 Επίση θα βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα μας. Ε, στο δεδομένο οικονομικό πλαίσιο ένας νέος ε, προπολογισμό θα πρέπει να χορηγεί περισσότερους πόρους στον τομέα της έρευνας, την κατάρτιση για τις πράσινες τεχνολογίες και η δημοσιονομική υπευθυνότητα για όπως ε, και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης πάνε χέρι-χέρι. Δεύτερη προτεραιότητα να υπάρξει μεγέθυνση, οικονομική μεγέθυνση της Ευρώπης. Το 2012 είναι, αποτελεί την 20η επέτειο από την έναρξη της ενίας αγοράς και είναι μία, ένα από τα σημαντικά, σημαντικότερα επιτεύγματα. Αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλο το δυναμικό που μας προσφέρει η ενία αγορά και η Ιδανική Προεδρία προτίθεται να ε, εργαστεί από αυτού. Τώρα, πράσινη Ευρώπη, τρίτο είναι προτεραιότητα. Θέλουμε να έχουμε μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση της πράσινης ε, ανάπτυξης. Οι ε, ε, ευρωπαϊκές οικονομίες θα πρέπει να γίνουν βιώσιμες πρόθεσμα. Έχουμε αναπτύξει μια σφαιρική πολιτική και έφτασε η ώρα να επιταχύνουμε αυτήν την πολιτική, μια οικονομική πολιτική όπου η οικονομική ανάπτυξη αποσυνδέεται από την ε, ανεξέλεγκτη χρήση των ε, πόρων και, το, και της ε, κατανάλωσης ενέργειας. τέταρτη προτεραιότητα μια ασφαλέστερη Ευρώπη, η ιδανική προεδρία θα ηγηθεί πολλών πρωτοβουλειών στον τομέα της δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. απαιτείται να ε, αποκτήσουμε ένα ενιαίο σύστημα χορήγησης ασύλου. Η Ιδανική Προεδρία θα φροντίσει να προωθήσει ένα ε, αποτελεσματικό σύστημα χορήγησης ασύλου σύμφωνα με το κεκτημένο του Σέγγεν. Ε, και σε αυτό που συζητόμαστε στην Καθρινάστον ε, και στην Επιτροπή εξωτερική Δράσης. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε την κυρία Άστον και την Επιτροπή εξωτερική Δράσης. Θα θέλαμε να αποτελέσουμε μια προεδρία μοντέλο για την ε, ευρύτερη συνεργασία με την Υπηρεσία εξωτερική δράση. Θέλουμε επίση να δραματίσουμε ενεργό ρόλο στην περιφέρεια και εδώ φτάνω στο θέμα της διεύρυνσης και την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία. Η πολιτική μας, ε, η πολιτική της διεύρυνσης είναι μία από τις πιο επιτυχημένες πολιτικές μας. Πρόκειται για μια πολιτική που στηρίζεται στο ε, θέμα της ε, προσθετικότητας και όλα αυτά με βάση την ευημερία και την ανάπτυξη του συνόλου της Ευρώπης σε περίοδο κρίσης. Βλέπω ότι η ελκυστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει άφεκτη. Ε, με το παράδειγμα αυτή της εβδομάδα στην Κροατία, όπου η συντριχή πλειοψηφία των ψηφισάντων ενέκριναν την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Επίσης, την διεύρυνση θεωρώ ότι θα πρέπει να, να διατηρήσουμε έναν, ένα διάλογο με το Κοινοβούλιο. Σημαντική προσφορά του Κοινοβουλίου θα είναι η εργασία των εισηγητών του Κοινοβουλίου με τις ε, χώρες που θέλουν μια στενότερη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτές οι εκθέσεις και η αφαίρεσή του στην Ολομέλεια θα αποτελέσει μια πολύ σημαντική συμβολή στις στρατηγικές συζητήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διεύρυνση. Επίσης πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο με, στο διάλογο με τις ενδιαφερόμενες χώρες θα συμβάλλει θετικά και σημαντικά για την καλύτερη κατανόηση του πώς λειτουργεί η Ευρώπη και ποια είναι ποιες αξίες βασιζόμεθα ως Προεδρία θα προωθήσουμε τον, ε, την ε, προσέγγιση βήμα προς βήμα. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου θέτουν ε, τη βάση για την επίλυση αυτών των ζητημάτων. Τώρα θα αναφερθώ στις επιμέρους περιοχές και κράτη. Η ευρωπαϊκή προοπτική είναι ένα πλαίσιο το οποίο μπορούμε να διασφαλίσουμε την επικοδομητική συνύπαρξη στην περιοχή ε, έχουμε εντολή αύριο στα λίγο κρατών και κυβερνήσεων να εξετάσουμε το ζήτημα του καθεστώτος υποψήφιας χώρας στη Σερβία. Η Σερβία έχει κάνει σημαντική πρόοδο και για να πληρεί τα πολιτικά κριτήρια και είναι πολύ ικανοποιητική η πρόοδος της ε, Σερβία επίσης έχει ε, συμμετάσχει στον διάλογο Βελιγραδίου Πριστίνας. Ε, θα χωρίς να διαπιστώσουμε ότι η Σερβία συνεχίζει να εφαρμόζει καλή την πίστη την συμφωνία που έχει συμπεριληφθεί στον διάλογο Πρίστινα Βελιγραδίου και τη συνεργασία με την K4 και την EULEX. Γνωρίζω πως ε, είχατε συζήτηση με τον Δανό Υπουργό Εξωτερικών ε, ειδικά επί συγκεκριμένων ζητημάτων και δεν θα αναφερθώ εξαντλητικά σε αυτά. Για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Μαύρο Βούνιο τον Ιούνιο, θα εξετάσουμε την πρόοδο του Μαυροβουνίου και θα ε, εστιάσουμε στο θέμα του ε, καταπολέμησης του οργανωμένου κλίματος, της διαφθοράς και του κράτος δικαίου. Ε, σημαντικά προσπάθειες θα καταβάλουμε για να, ε, να μπορέσουν οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να πληρώσουν τις ε, υποχρεώσει τους ε, τώρα σε ό,τι φορά την Τουρκία. Ελπίζουμε σε μια συνέχιση των διαπραγματεύσεων ε, για τη διεύρυνση. Πιστεύουμε ότι είναι προς το συμφέρον μας να διατηρήσουμε την Τουρκία στην ευρωπαϊκή πορεία. Γνωρίζετε ότι οι διαπραγματεύσει δεν προχωρούν με γοργοβήμα, αλλά εξετάζουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν και οποιαδήποτε ευκαιρία για πρόοδο θα την δράξουμε. Θέλουμε να υποστηρίξουμε την προτάσεις της Κομισιόν για μια θετική ατζέντα. Η ατζέντα αυτή έχει εξεταστεί από κοινού με την τουρκική πλευρά, αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτή η ατζέντα θα είναι συμπληρωματική ε, των διαδικασιών διεύρυνσης. Να αναφερθώ επίσης στην Ισλανδία. Οι διαπραγματεύσεις ε, έχουν προχωρήσει και ε, η Ισλανδία είναι μια χώρα υποψήφη σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο 23. Ε, θα έλεγα ότι το ανοίξαμε και το κλείσαμε ε, ταυτόχρονα. Η Ισλανδία θα πρέπει να πληρεί τα ίδια κριτήρια όπως και οι υπόλοιπε υποψήφιε χώρες. Τα θέματα που με την ε, Ισλανδία άπτονται τον ε, της αλίας. Μερικά είναι πιο περίπλοκα από άλλα, αλλά πιστεύουμε ότι θα προχωρήσουμε τις διαπραγματεύσεις ε, ανοίγοντας και κλείνοντας σημαντικά κεφάλαια κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Επίσης θα ήθελα να πω μερικά λόγια για την πολιτική γειτονία. Είναι σημαντική. Η πολιτική γειτονία θα πρέπει να συνεχίσει την ε, προσέγγιση που είχε ακολουθήσει μέχρι τώρα. Θέλουμε να, να προωθήσουμε με τους γείτονές μας ε, οικονομική συνεργασία, πολιτική ολοκλήρωση και ε, δημοσιοοικονομική βοήθεια. Η Κομισιόν και η Ιδανική Προεδρία θα εργαστούν για την αναθεωρημένη πολιτική της ε, γειτονίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα καταβάλουμε προσπάθειες ε, για πρόθεση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα πρέπει οι εταίροι μας ε, να γνωρίζουν ότι μπορούν να στηρίζονται πάνω μας ό,τι φορά την ε, ανατολική διάσταση και εταιρική σχέση έχουμε προχωρήσει στις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και οι διαπραγματεύσεις προχωρούν με την Μολδαβία, την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και την Γεωργία. Αρνητικές εξελίξεις στην Λευκορωσία κατέστησαν αδύνατον να υπάρξει παρόμοια συνεργασία όπως με τις υπόλοιπες χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. Φυσικά παρακολουθούμε την κατάσταση στην Ουκρανία από κοντά και ελπίζουμε ότι οι ε, αλλαγές στην εσωτερική πολιτική θα καταστήσουν ε, δυνατόν να υπογραφεί η Συμφωνία Σύνδεσης. Όταν πρόκειται, μιλάμε για την Συμφωνία Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, σε συνεργασία με την Κομισιόν θα προετοιμάσουμε έναν χάρτη πορείας. χάρτης πορείας θα εξεταστεί το Μάιο-Ιούνιο στην Υπουργική Διάσκεψη ε, και θα ενημερώσω φυσικά ε, τους εταίρους μας εγκαίρους τώρα για τους ε, εταίρους μας του Νότου ε, υπόθηκαν πολλά, αλλά θα επαναλάβω μερικά πράγματα. Η Αραβική Άνοιξη μα προσφέρει μια ιστορική πρόκληση στην Ευρώπη. Ε, η συνθήκη της Λισαβόνας ε, μας έδωσε νέες ε, εξουσίες στην, εξωτερική πολιτική. Έχουμε ενδιαφέρον πολύ σημαντικό για μια στα, σταθερές δημοκρατίες στην περιοχή και μια περαιτέρω απελευθέρωση των οικονομίων της ναι, φυσικά υπάρχουν ανησυχίε από πλευρά ε, βιομηχανιών που πλήττονται από κάποια μέτρα, αλλά και αυτέ οι ανησυχίε δεν πρέπει να παραμεληθούν, δεν πρέπει να ξεχνάμε το βασικό στρατηγικό μας ε, συμφέρον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας ε, φυσικός εταίρο της ε, Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής. Μερικά λόγια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως ε, ζητήθηκε από την Επιτροπή σας. πράγωγη για προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεμελιώδων ελευθεριών, δημοκρατία και κράτου δικαίου. Είναι οι ε, θεμελιώδει αρχέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτέ οι θεμελιώδει αρχέ κατευθύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι κράτη τη τόσο στο εσωτερικό τη όσο και προ το εξωτερικό. Όπως ε, δήλωσε και είπε εκπρόσωπος στις 13 ε, Δεκεμβρίου εδώ ενώπιον του Κοινοβουλίου. Η Ιδανική Προεδρία θα μπορεί πάρα να συμφωνήσει απόλυτα με τα λόγια της ε, κυρίας των το ζήτημα αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο τη υπηρεσία εξωτερική δράση. Ε, η Ιδανική Προεδρία καλωσορίζει τι προτάσει για δράση που συμπεριλαμβάνονται στο πλαίσιο τη ανακοίνωσης ε, και μιλάμε για την ε, δημιουργία εταιρικών σχέσεων και μα ζητείτε να μιλήσουμε με μία φωνή. Με μία φωνή 27 κράτη-μέλη, όπω καταλαβαίνετε, έχουν πολύ μεγαλύτερο απόϊχο οι περιθήκες δράσεις ε, είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την υλοποίηση των ε, στόχων της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε. Πέρυσι είχαμε πολλά παραδείγματα αναφορικά με τον οικουμενικό χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε συνδυασμό με την Αραβική Άνοιξη υπήρξε ε, έχουμε την ε, Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που φέτος ε, συμπληρώνει 60 έτη. Επίση, προσβλέπουμε σε μια στενή συνεργασία με την Επιτροπή σας. μοιραζόμαστε τις ίδιε αξίες, τα ίδια καθήκοντα και τώρα θα πρέπει να κάτσουμε και να δουλέψουμε σκληρά. Ευχαριστώ για αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα εργασίας. Ελπίζω να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε να πετύχουμε επικοδομητικά αποτελέσματα. Ο κ. Κασουλίδης και όλοι όσοι μιλήσουν ένα λεπτό, γιατί εννέα ομιλητές έχουν ζητήσει το λόγο. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ καλωσορίζω τον Υπουργό και του εύχομαι και εκείνον και στη χώρα του επιτυχή Προεδρία έτσι ώστε τα αποτελέσματά της να να είναι θετικά και για την Κύπρο που θα αναλάβει την επόμενη Προεδρία και θα μπορέσει να βασιστεί σε εκείνα τα αποτελέσματα. Και οι τέσσερις προτεραιότητες που αναφέρατε αλλά και τα προγράμματα και τα σχέδια για την πολιτική γειτονία ανθρώπινα δικαιώματα και διεύρυνση μας ε, βρίσκουν σύμφωνους. Όσο για το ρόλο του Κοινοβουλίου σημειώνουμε μεγάλη ικανοποίηση ότι πράγματι στις προσπάθειες για διεύρυνση και ο αρμόδιος συζητητής και άλλοι συνάδελφοι μπορούν να σας βοηθήσουν ώστε πρώτα απ' όλα να προωθηθεί η ενταξιακή προοπτική των Βαλκανίων, δεύτερον η διεύρυνση προς την Τουρκία, γιατί όπως σας είπα και άλλες φορές, λένε ότι η Τουρκία θα αφαιρθεί με πολύ επαγγελματικό και ουδέτερο τρόπο κατά την Προεδρία της και θέλω να μπορέσετε εσείς προηγουμένως να πείσετε την Τουρκία να ανοίξει και τα επόμενα κεφάλαια Πράγμα που θα προσπαθήσει να κάνει και η Κύπρος. Χαίρομαι γιατί είπατε ότι το θετικό αυτό πρόγραμμα δεν υποκαθιστά τις ίδιες τις διαπραγματεύσεις. Και τώρα το ερώτημα για την πολιτική της γειτονίας. Θέλω να σχολιάσετε το θέμα των διωγμών χριστιανών που φοβάμαι ότι χειροτερεύουν στις χώρες που, όπου, έγινε οι αραβικές, όπου έγιναν οι αραβικές επαναστάσεις αλλά και στο Ιράκ. Εμείς οι Ευρωπαίοι είμαστε πολύ ευαίσθητοι σε θέματα ρατσισμού, ξενοφοβίας και δίωξης οποιασδήποτε θρησκείας. Σας ευχαριστώ. Αυτό ήταν δυόμιση λεπτά όμως. Ελπίζω ο σοσιαλιστής συντονιστής να φερθεί καλύτερα. Εγώ, εγώ είμαι πάντα πειθαρχημένος κύριε Πρόεδρε. Κύριε Βάμεν, σας ευχαριστώ που αναφέρατε τις προτεραιότητες σας, ειδικά το φιλόδοξο πρόγραμμά σας. Τα πάει καλά η Δανία με τις διευρύνσεις και είμαι σίγουρος πως και αυτή η Προεδρία θα αποτελέσει και πάλι θετικό παράδειγμα. Έχετε την ευκαιρία να, καθαστη, να καταστήσετε πλέον ε, αναπόδραστη την ε, διεύρυνση των Δυτικών Βαλκανίων με το να γίνει η Σερβία ε, υποψήφια χώρα. Ε, τέλος πάντων είναι ένα δύσκολο ζήτημα αυτό που πρέπει να αντιμετωπιστεί τη Τουρκία δηλαδή σε Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και τα έχετε τη στήριξη του Κοινοβουλίου και τα εξωτερικά μέσα βεβαίω, ειδικά την προενταξιακή βοήθεια και είμαι σίγουρος πως μπορούμε να συνεργαστούμε ε, μέχρι το τέλος της Προεδρίας σας. Μια σύντομη παρατήρηση για την πολιτική γειτονία. Υπάρχουν διάφορες εκλογικές αναμετρήσεις. Αναφέρατε τη Ρωσία και υπάρχει Λευκορωσία, ε, Ουκρανία και πιθανώς και η Μολδαβία γιατί βλέπουμε αρνητικές εξελίξεις σε κάποιες χώρες πρέπει να είμαστε προσεκτικοί δεν θα πρέπει και οι υπόλοιποι να ξεφύγουν από το δρόμο την πορεία τους τέλος πρέπει να λάβουμε υπόψη πως και η Ρωσία με την ιδέα αυτή του Πούτιν της Ευρασιατικής Ένωσης βλέπουμε πως υπάρχει μια θετική υποδοχή αυτής της ε, ιδέας στις χώρες αυτής της Ανατολικής Γειτονίας. Υπάρχει προπαγάνδα ρωσική, πρέπει να είμαστε λοιπόν πάρα πολύ προσεκτικοί για τις ε, εξελίξεις αυτές. Ευχαριστώ. Ε, ήμουν πιο πειθαρχημένο σε πάση περιπτώσει από τον συνάδελφο κύριε Πρόεδρε. Το πρόεδρος χωρίς μικρόφωνο. Ε, τουλάχιστον λίγο παραπάνω. Λίγο πιο πειθαρχημένος απαντάει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα εξ ονόματος των να καλωσορίσω βεβαίω ε, την προσήλωση του κυρίου Υπουργού στη διεύρυνση, αλλά θέλω να ρωτήσω κάποια πράγματα. Πρώτον, δουλειές και ανάπτυξη. Κύριε Υπουργέ, βλέπετε πιθανότητα διεύρυνσης της ε, ενιαίας αγοράς. Τι θα κάνετε ιδιαίτερα για να προτρέψετε την Κομισιόν για να ανοίξει η ενιαία αγορά υπηρεσιών που θα προσθέσει οπωσδήποτε σε δουλειά και ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, για το πράσινο πρόγραμμά σα με τους συναδέλφους σα στο Συμβούλιο θα υιοθετήσετε τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού ιδρύματο Κλίματος. Ένα οδικό χάρτη για το 2050 που μας λέει πώς θα πάμε ε, από εκεί που είμαστε σήμερα στο που πρέπει να πάμε στο 2050 για να κοπούν οι εκπομπές κατά 80%. Uh, Δύο ερωτήσεις ε, έχω εγώ. Θεωρείτε πως έχετε την παραμικρή πιθανότητα να επιτύχετε συμφωνία για τα μέσα επίλυσης της οικονομικής κρίσης, είτε είστε εντός είτε εκτός Ευρωζώνης. Και δεύτερον, δεδομένη της ε, εμπειρίας της Δανίας για επιθέσεις στην ελευθερία των ΜΜΕ, τι σκοπεύετε να κάνετε για να προστατεύσετε αυτή την ε, θεμελιώδη δημοκρατική ελευθερία. Αν εγώ μπορώ να μιλήσω ένα λεπτό, τόσο μπορούν και άλλοι νομίζω. Edit. Τελευταίος γι' αυτό το γύρο, η κυρία Κοντούρη. Minister. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον Υπουργό. Έχετε πολλές προκλήσεις, κάτι το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Αναφέρατε κάποια σχόλια που υπήρξαν στον τύπο της Δανίας για το ότι είναι δύσκολο το Κοινοβούλιο και να συνεργαστεί κανείς με το Κοινοβούλιο. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τα σχόλια αυτά. Κύριε Υπουργέ. Uh, Ευχαριστώ και να ξεκινήσω λέγοντας ε, πως χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δίνετε ευκαιρία να απαντήσω σε ερωτήσεις σας και τα σχόλια σας. Προς τον κύριο Κασουλίδη. Η Κύπρος ε, θα κάνει μια προεδρία σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πω ότι από τη Ιδανική Προεδρία. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην, ε, στην Κυπριακή Σύνομη που θα μας διαδεχθεί και το βλέπουμε σε μια περαιτέρω συνεργασία. Ο κύριος Κασουλίδης ε, έστειξε επίσης ε, το ζήτημα των χριστιανών στην Βόρειο Αφρική. Είναι πάγια θέση της Δανικής Προεδρίας αλλά και όλων των μελών του Κοινοβουλίου ότι θα προστατεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και το δικαίωμα στην ανεξιθρησκεία, στην ελεύθερη λατρεία. Γι' αυτό λοιπόν αν επιθέσεις γίνουν κατά των χριστιανών, φυσικά και μας ανησυχεί το ζήτημα, είναι κάτι που θα πρέπει να το εξετάσουμε εάν τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Σχετικά με την ερώτηση του κυρίου Βίγκενιν από τη Βουλγαρία, ο οποίος δήλωσε πως αναπόδρεπτα βήματα μπορούν να αναλυφθούν κατά, για το, την Ιντανική Προεδρία ε, στο, ε, για τη Σερβία και το Μαυροβούνι Ελπίζω ότι η λύση μπορεί να εξευρεθεί στο σερβικό ζήτημα, στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων το Φεβρουάριο και μετά από έγκριση από το Συμβούλιο τον Μάρτιο, όπως ακούσατε από τον ε, Υπουργό Εξωτερικών, η διαδικασία πάει προς την κατεύθυνση, αλλά πρέπει κάποια πράγματα να εξεταστούν περαιτέρω. Ελπίζουμε ότι και το Μαυροβούνιο θα ακολουθήσει την ε, πρέβουσα οδό. Τώρα, για την ε, Θήρομ, για την πρώην Ιουκλαβική Δημοκρατία Μακεδονίας, ε, έχουμε καταστήσει σαφές σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ότι θέλουμε να εξευρεθεί λύση και αυτό θεωρούμε ότι είναι προς όφελος όλων των εμπλεκομένων, προς όφελος όλων και πιστεύουμε ότι αυτό θα συμβεί. Ξέρουμε ότι το ζήτημα είναι δύσκολο αλλά απαιτείται λύση και η λύση θα πρέπει να βρεθεί από τα ενδιαφερόμενα μέρη και ζητήσαμε από τα ενδιαφερόμενα μέρη να το πράξουν. Ο κύριος Βότσον είπε πώς μπορούμε να κάνουμε περισσότερο για την απασχόληση και την ανάπτυξη. Τα θέλαμε η αγορά να προωθήσει τις 12 ε, δραστηριότητε της ε, Κομισιόν, της Πρωτοβουλίας Κομισιόν και είμαστε πεπισμένοι πως και το Κοινοβούλιο το αυτό θα πράξει. Θα είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την ε, περαιτέρω ανάπτυξη την οικονομική στην Ευρώπη και ότι και σε αυτό θα συμβάλλει φυσικά και το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο κύριος Άτκινς είπε, ρώτησε μάλλον, αν η Δανία έχει κάποια επιρροή σε θέματα οικονομικών θα κάνουμε ό,τι μπορούμε κατά διάρκεια του δανεικού εξαμήνου Ξέρουμε ότι οι διαπραγματεύσει συνεχίζονται σε πολλούς τομείς και εμείς θέλουμε να αποτελέσουμε γέφυρα ανάμεσα στου 17 τη Ευρωζώνη και τους υπολείπου 10. Επίσης θα μιλήσουμε για τις δημοκρατικές αξίες όταν μιλήσουμε για την ελευθερία τύπου όπως υπόθηκε. Αυτό είναι σημαντικό και για την Δανική Προεδρία αλλά και για τη Δανία γενικότερα τέλος ε, Γκρούμπεργκ από την Φιλανδία είπε ότι θα ρώτησε μάλλον θα είναι σημαντικό να εργαστούμε με το Κοινοβούλιο. Ναι, φυσικά, εμείς δεν θέλουμε να είμαστε μόνο λόγια. Ελπίζουμε, ε, μάλλον ότι το Κοινοβούλιο θα είναι ένας ε, εταίρος υψής της σημασίας και σοβαρότητας όταν έχουμε για παράδειγμα τη μετέθμιση της ενίας αγοράς όπως είπα και στις εισαγωγές παρατηρήσεις θεωρούμε ότι οι εισηγητές μπορούν να δεματίσουν ένα σημαντικότατο ρόλο και εμείς θα τίνουμε δίκο νους σε αυτούς τους εισηγητές του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Thank you, Minister. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Δεύτερος γύρος, ο Κόμις του Ντάρνης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, αρχίσατε μιλώντας για την οικονομική διακυβέρνηση, governance, και μετά μιλήσατε για ανθρώπινα δικαιώματα που σωστά τα ονομάσατε πανανθρώπινα. Αλλά οι επιπτώσεις της συμφωνίας αυτής για τη διακυβέρνηση μπορεί να είναι δημοψήφισμα στην Ιρλανδία. Ερωτώ λοιπόν. Η ιδανική προεδρία προτίθεται να σεβαστεί και να δεχτεί το αποτέλεσμα ενός τέτοιου δημοψηφίσματος στην Ιρλανδία για τη συμφωνία ή συνθήκη αυτή ή μήπως τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν εφαρμόζονται όταν δεν βολεύουν όπως έκαναν οι προκάτοχοί σας. Ευχαριστώ κυρία Γκόμες. Μιλήσατε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στην οικονομική πλευρά. Κοιτάξτε, εγώ θα αναφερθώ και στις αναποτελεσματικές πολιτικές οι οποίες ε, έδωσαν τροφή στην κερδοσκοπία. Η Προεδρία λοιπόν της Δανίας θα ζητήσει από τους υπουργούς να ασχοληθούν με τις συνέπειες που έχει αυτό στα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ΚΕΠΑ και την ε, κοινή εξωτερική πολιτική. Δείτε την Πορτογαλία, τη χώρα μου, όπου οι λεγόμενες ιδιωτικοποίησεις τι έκαναν, έδωσαν στρατηγικά ε, μερίδια στην ε, ΔΕΗ και στο εθνικό δίκτυο. Σε ποιον, στο εθνικό, στο ε, σε κινέζικη εταιρεία, δηλαδή στο Κινέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα που ελέγχει την εταιρεία. Οι συνέπειες είναι τρομερές. Αυτό συμβαίνει και σε προωθημένη τεχνολογία στον τομέα της άμυνας. Θα αναγκάσετε τους υπουργούς να σκεφτούν το τι σημαίνει αυτό για την πολιτική διεύρυνση και την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Ευχαριστώ κύριος Κούκαν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, ξεκινήσατε λέγοντα πω η πολιτική διεύνηση είναι επιτυχημένη πολιτική τη Ένωση. Νομίζω πρέπει να την αναπτύξουμε και να έχουμε την ίδια προσέγγιση και στο μέλλον. Ήσασταν πολύ λεπτομερεί. σε χώρες όσον αφορά όπως η Σερβία, Μαυροβούνιο, Πογοδομού, η Ισλανδία. Α, δεν είναι πρόβλημα, αλλά Οπωσδήποτε οι αποφάσεις που αναβλήθηκαν από πέρσι θα πρέπει να ληφθούν ε, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πως υπάρχουν και άλλες χώρες που θα θέλαμε να κρατήσουμε στην ευρωπαϊκή πορεία. Η Αλβανία μετά από, ε, πολιτική, μετά από ένα πολιτικό τέλμα έχει επιτέλους σωτικές ειδήσεις. Η Βοσνία Αρζεγοβίνη είναι δύσκολη περίπτωση αλλά κάποιο αποτέλεσμα επιτέφθη. Επίσης για το κοσυφοπαίδιο, απελευθέρωση θεωρήσεων και διάλογο οι χώρες αυτές όταν κάνουν κάτι σωστό νομίζω πως πρέπει να τις επιβραδύνουμε. Δεν πρέπει να τις ξεχνάμε. Έχετε λοιπόν ε, μπροστά σας δύσκολη δουλειά και εύχομαι καλή τύχη. Ευχαριστώ η κυρία Μπουσκούρτ τελευταία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. έχετε μία θετική ατζέντα όσον αφορά την Τουρκία. Γιατί ε, δεν έχουμε ξανακούσει τίποτα από την προηγούμενη Προεδρία και μετά. Θα κάνετε κάτι τίποτα επιτέλους. Ναι. δεύτερον, η Βοσνία και η μετά από ένα χρόνο διαπραγματεύσεων απέκτησε κυβέρνηση. θα βοηθήσετε για να προωθηθεί και αυτή η χώρα. Τελευταία ερώτηση. Εγώ σας γνώρισα σε μια συνάντηση που είχαμε για τα δικαιώματα των γυναικών με τις σοσιαλίστριες. Το ερώτημά μου είναι, στην πολιτική γειτονία, Βόρεια Αφρική, Αραβικές χώρες και τα λοιπά, πόσο θα θίξετε το θέμα των δικαιωμάτων των γυναικών. Σας ευχαριστώ κυρία Μποσκούρτ. Τώρα, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Θα σας κατευχαριστώ. Πρώτον, ο κόμις του Ντάρτμουθ. Σέβομαι απολύτως οποιοδήποτε αποτέλεσμα θα, θα καταλήξουν οι Ιρλανδοί πολίτες. Έχουν φυσικά τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους, ιδίως ανθρώπινα. Αυτή είναι η θέση της Δανικής Προεδρίας και ελπίζω και όλων των υπολείπων Προεδριών. Θα συνεργαστώ με τους Ιρλανδούς που θα έχουν την Προεδρία μετά την Κύπρο. Και είμαι βέβαιος ότι και η Ιρλανδία θα παίξει σημαντικό ρόλο στην οικογένειά μας. Για την κυρία Γκόμες τώρα είπε ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι μεταρρυθμίσεις και οι πρωτοβουλίες των χωρών μελών έχουν επιπτώσεις και καμιά φορά επιπτώσεις απρόβλεπτες. Νομίζω ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς και επίσης ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση, όχι μόνο της Πορτογαλίας αλλά οποιοδήποτε χώρα μέλους, έχει δικαίωμα να πάρει σκληρές αποφάσεις, αλλά πρέπει να το κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να διασφαλίσει τα συμφέροντα της χώρας της. Αυτό τελικά είναι η ευθύνη κάθε κυβέρνησης και όχι ειδικά της Δανικής Προεδρίας. Παρέμβαση χωρίς μικρόφωνο. Συμφωνώ. Συμφωνώ κύρια ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολύ δύσκολη περίοδο της ιστορίας του, της, και ότι τα κράτη-μέλη παίρνουν δύσκολες αποφάσεις και το καθένα, οι αποφάσεις του καθενός επηρεάζουν και τους άλλους, έχουν επιπτώσεις και στους άλλους. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι είναι θέμα κυριαρχίας του κάθε κράτους και κυβέρνησης να επιλέξει το καταλληλότερο εργαλείο για τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόσει τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Μπορεί κανείς να συμφωνεί ή να διαφωνεί ανάλογα με την πολιτική του φιλοσοφία, αλλά δικαίωμα της κάθε χώρας είναι να πάρει την απόφαση αυτή. Ο κύριος Κούκαν είπε ότι συμφωνεί ότι είναι σημαντικό να μιλήσουμε για τα Βαλκάνια και την ανάπτυξή τους αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι χώρες αυτές δεν θα ζητηθούν μόνο τον Μάρτιο και ότι υπάρχουν και άλλες χώρες που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Για την Αλβανία χαιρετίζω τη συνεργασία μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και τη δημιουργία μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής για τις εκλογικές μεταρρυθμίσεις. Αλλά και μετά την απόφαση στη λεγόμενη υπόθεση ΜΙΤΑ που εξέπληξε πολλούς, είναι σημαντικό να υπάρξει σημαντική πρόοδος για την επιβολή της τάξεως για τη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη που ανέφερε η κυρία Μποσκούρτ Χαίρομαι γιατί έχει υπάρξει εκεί μια συμφωνία και αναμένω την έγκριση και της κυβέρνησης. Για τις βασικές μεταρρυθμίσεις περιμένουμε περισσότερη ε, πρόοδο, αλλά βασικά θα ήθελα να πω ότι οι χώρες που αναφέρατε θα ήθελα να έχουν μακροχρόνιες προοπτικές για ένταξη του, της δημοκρατικής μας, στη δημοκρατική μας λέσχη. Υπάρχει όμως πολλής δρόμος ακόμα. Μετά ακούστηκε μια ερώτηση επίσης για, α, για την Τουρκία. Για την Τουρκία της ίδιας κυρίας Μποσκιούρτ. Αν αναμένουμε δηλαδή να ανοίξουν νέα κεφάλαια στις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία αν γίνεται γιατί όχι. Αλλά δεν αναμένω και θαύματα για τις διαπραγματεύσεις αυτές με την Τουρκία γιατί όλοι γνωρίζουν ότι είναι πολύ δύσκολες. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αλλά, αλλά ο Καρσιλαμάς χρειάζεται δύο. Έχουμε πολύ σκληρή διαπραγμάτευση μπροστά μας και ξέρουμε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα για το τουρκικό θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Μόλις τελειώσαμε ακριβώς 6.30. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και σας εύχομαι εξ ονόματός μου και της Επιτροπής μας καλή επιτυχία στη Δανική Προεδρία. Τελειώσαμε τη συνεδρίαση, η επόμενη θα είναι την Τρίτη στις 31 Ιανουαρίου στις 10 το πρωί. Ευχαριστώ πολύ, Καληνύχτα.